Να αρχίσουμε, συνάδελφοι, γιατί έχουμε πολλά θέματα στην ημέρα στη διάταξη, λέει ο Οπότε το ένα το κάναμε, ε, ξεκινήσαμε δηλαδή με την συνεδρίαση των συντονιστών και πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 2, που είναι η έγκριση της ημέρας της διάταξης. Ε, υπάρχει μία διορθωσούλα που πρέπει να γίνει και ε, είναι ο τίτλος του καλεσμένου μα για το 17 όσον αφορά την ολοκληρωμένη απάντηση στο ζήτημα των προσφύγων και ο σωστό τίτλο για τον φιλοξενούμενό μα, τον Μαμαντού Νταν Μπάλντε, είναι αναπληρωτή διευθυντή ε, του, του μήματο τη υπηρεσία τέλο πάντων για την ε, αντοχή, ανθεκτικότητα και τι λύσει τη της ΥΠΑ του για τους πρόσφυγες και κάποιες ανακοινώσεις τώρα πρώτα πρώτα στην τελευταία μας συνάντηση Είχαμε επικοινωνήσει μέσω του Skype με τον κύριο Warden συγγνώμη, από τον, ε, τον επικεφαλής του Εθνικού Πάρκου Βιρούγκα με τον πρίγκιπα ε, Εμμανουήλ όσον αφορά κάποιο είδους ε, εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί εκεί ένας οδηγός, ε, πέντε φύλακες είχαν ε, φωνευτεί, ε, απαγωγές και λοιπά, όλα αυτά υποσκοτεινές συνθήκες και δεν ξέρω η κατάσταση εκεί πέρα έχει επιδεινωθεί και στο Κονγκό και επίσης έχουμε στις εκλογές τις 23ης του 10 που δεν ξέρουμε αν θα γίνουν και επίσης υπάρχουν διάφορα προβλήματα εκεί πάρα πολλοί φεύγουν και για λόγους δημόσιας υγείας περνάνε από το Κονγκό στην ε, Ουγκάντα και επίσης ε, ε, από τις 8 Μαΐου επισήμως η χώρα έχει κηρυχθεί κατάσταση αγερμού λόγω του ιού έμπολα και αυτό επίσης πρόκειται να επηρεάσει την κατάσταση οπότε αφού υπάρχει αυτό το ξέσπασμα και αυτό μπορεί να γίνει στις γειτονικέ χώρες όπως έγινε και στη Δυτική Αφρική και αυτό μπορεί να πάει εκεί που υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγες και πάρα πολλοί φτωχοί Οπότε θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την κατάσταση στη Δημοκρατία του Κονγκό από κοντά τους αμέσως μήνες. Ε, όπως ξέρετε θα έχουμε τις ημερίδες για την ε, ε, ανάπτυξη από πλευράς της Ευρώπης 5 και 6 Ιουνίου όποιος ευρωβουλευτής ή κάποιος συνάδελφος δηλώσει να πάει ε, πρέπει να απευθυνθεί στην ε, γραμματεία, μπορεί να το κάνει και ιντερνετικά υπάρχει όμως προθεσμία 18 Μαΐου αν θέλετε να πάτε σε αυτές τις Ευρωπαϊκές Ανάπτυξης τώρα μέχρι την Παρασκευή να το δηλώσετε και επίσης όσον αφορά τους γάμους ανηλίκων θα έχουμε κάποια εκδήλωση από εμείς η Επιτροπή μας και ο Σαρλ Γκιόρενς πρόκειται να διευθύνει το σχετικό πάνελ θα έχουμε από Νίγερα και Μπαγκλαντές ε, κάποιους ε, ανηλίκους Τετάρτη 6 Ιουνίου 11.30 με 1 Επομένως, αν θέλετε να πάτε σε αυτές τις μερίδες ανάπτυξης, να το δηλώστε. 5 και 6 Ιουνίου. Τώρα, το υπαριθμό 4. Έγκριση των πρακτικών να τα έχετε λάβει στο φάκελο. Αν υπάρχουν παρατηρήσεις να τα πείτε στην γραμματεία πριν το τέλος της συνεδρίασης και αν δεν υπάρχουν ενστάσεις θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται 5 αποφάσεις συντονιστών και συστάσεις της 24ης ε, και αυτά να τα πείτε αν έχετε αντίρρηση ή στην γραμματεία αλλιώς θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται ανακοινώσει από την Επιτροπή. Θα έρθουν δύο επίτροποι. Αυτά για τις ανακοινώσει. Εφτά. Ε, αναπτυξιακή χρηματοδότηση. Ε, τηρούν τις δεσμεύσεις τους η Ένωση και τα κράτη-μέλη. Και όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σταμάτησε τις εκθέσεις ή αναφορές τέλος πάντων λογοδοσίας ε, αυτό ήταν κάτι το, το οποίο θέλησαμε αρνητικό και είναι το θέμα αυτού του στόχου 0,7% οπότε και είπαμε ε, να έρθει η Επιτροπή να τα συζητήσουμε τα σχετικά με τις επενδύσεις της βιώσιμης ανάπτυξης ε, όπως τα ανέθεσε, όπως, συγγνώμη, όπως τα ανέπτυξε ο κύριος Μίμητσος στη Νέα Υόρκη. Ήρθε τώρα εδώ ο κύριος ε, Σαραζέν να μας τα πει. Να δούμε πού βρισκόμαστε, πού τα πάμε καλά και πού δεν τα πάμε καλά όσον αφορά τις υποσχέσεις μας. Το 2015 δεν πετύχαμε τον στόχο του 0,7 και δώσαμε τώρα παράταση 15 ετών για να πετύχουμε αυτό το 0,7%. Έχουμε μπροστά μας χρόνο γιατί είμαστε μόλις το 2018. Οπότε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σαραζά. Καλώς όρισαν ε, οι Γερμανοί διδάσκαλοι τους οποίους έχουμε δώσει, φιλοξενουμένους, είναι πίσω-πίσω. Ο Νόρμπετ Νόζερ τους έχει καλέσει, βρίσκονται στο βάθος αιθούσης. Ενδιαφέρεσε, ενδιαφέρεστε για την βιώσιμη ανάπτυξη σε επίπεδο σχολείων, σε επίπεδο στόχων. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό γιατί έτσι οι νέοι συμμετέχουν στην προσπάθεια για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και τα παιδιά μπορούν να μεταδώσουν ε, ε, το, το, το μήνυμα στους ε, γονείς τους. Και άλλωστε αυτά τα παιδιά, οι μαθητές, το 2030 θα είναι ενήλικοι. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ένα χειροκρότημα για τους Γερμανούς δασκάλους. Okay, so colleagues... Ωραία. Συνόδελφοι, έχετε λάβει τη σχετική έκθεση για τι επενδύσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Και θα δώσουμε τώρα τις κοιτάξει του κύριο Σαραζέν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω τη χαρά λοιπόν να σας παρουσιάσω την έκθεση αυτή. Στην έκθεση περιγράφονται τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα στο 2015 και 2017 για την επίτευξη των στόχων τη θεματολογίου της Αντίσα Η προηγούμενη έκθεση λογοδοσίας ε, ήταν διαφορετική, τώρα η δομή έχει αλλάξει έτσι ώστε να συμφωνεί με το θεματολόγιο της Αντίσα Έτσι λοιπόν αποτελείται από πολλά τμήματα και από πολλούς τομείς δράσης. Εστιάζει ειδικότερα στις ε, προτεραιότητες σχετικά με την ε, συνένεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται για πρώτη φορά ε, συστήματα φωτεινού σηματοδότη τα οποία χρώματα αντιστοιχούν με, την, με το επίπεδο επίτευξης των στόχων από τα επιμέρους κράτη-μέλη. Αξιολογείται η προσπάθεια διότι αυτό είναι και ο κύριος θεματικός άξονας της έκθεσης. Πέραν της προόδου υπάρχει και ένας δεύτερος δείκτης για τους επιμέρους σχετικούς στόχους, διότι πολλές φορές οι στόχοι είναι αρκετά γενικοί για να μπορούμε να αξιολογήσουμε τις επιμέρους δράσεις στα κρατη Έτσι λοιπόν υπάρχει ο συγκεκριμένος δείκτης για το επίπεδο προσπάθειας. Σε γενικές γραμμές βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν ανταποκριθεί στους στόχους ε, του θεματολογίου με ίδιους πόρους και βρίσκονται στο σωστό δρόμο προς την επίτευξη των ε, στόχων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Εάν δούμε τώρα τα κεφάλαια ένα προς ένα, θα παρατηρήσουμε ότι σε ό,τι αφορά τους εγχώριους δημόσιους πόρους, τα κράτη-μέλη είναι οι κύριοι δωρητές για κεφάλαια κινητοποίησης και αύξησαν κατά πολύ τα κονδύλια για την κινητοποίηση των πόρων τα τελευταία δύο έτη. Σε ό,τι αφορά της ε, Διεθνής Δημόσιας και ιδιωτικές ε, χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, Διακόπτη Πρόεδρο, σε ποια σελίδα βρισκόμαστε στην έκθεση θα μας βοηθούσε, διότι δεν έχουμε την παρουσίασή σας και δεν μπορούμε να βρούμε αυτό στο οποίο αναφέρεστε. Ναι, αναφέρομαι στο κεφάλαιο 4, Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία, σελίδα 35 της έκθεσης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ζητήματα επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Στην έκθεση λοιπόν επιβεβαιώνεται ότι τα κράτη-μέλη παραμένουν ο μεγαλύτερος ε, πάροχος της επίσημης αναπτυξιακής ε, βοήθειας σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2017. Το 2017 τα επίπεδα φτάσαν στο 8,5% του ακαθάριστου ε, εθνικού προϊόντος. Σε σχέση με το 2016 όπου ήμασταν στο 0,53%. Το μόνο προβληματικό σημείο στην έκθεση αφορά την στασιμότητα. Βρισκόμαστε στο 0,11% του ΑΕΠ και στόχος είναι να φτάσουμε το 0,15% μέχρι το 2020 και το 0,20% μέχρι το 2030. Αυτό λοιπόν είναι το κύριο σημείο στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε και αναφέρεται στην έκθεση. Έπειτα. Σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε την πρόοδο σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Για παράδειγμα, βελτιώθηκε η επίδοση μας ε, στα, στις κοινέ δράσεις και στην εφαρμογή τους. Επίσης, είμαστε οι μεγαλύτεροι συνεισφέροντες στη χρηματοδότηση για το κλίμα. 22 δισεκατομμύρια δολάρια διατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν διαθέσει το 15% των παγκόσμιων υποχρεώσεών τους ε, στην ε, αναπτυξιακή συνεργασία. Ας περάσουμε τώρα στο κεφάλαιο 5, στην σελίδα 62 της έκθεσης. βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τα μέσα για το εμπόριο και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες έτσι ώστε να βοηθήσει τις χώρες αυτές να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις, στην αγορά. Και βλέπετε τα διάφορα μέσα που χρησιμοποιούνται. Ανάμεσα στο 2010 και το 2016 τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διπλασίασαν τις ε, δεσμεύσεις τους. Και αυξήθηκε η συμμετοχή στην ε, αγορά που αφορά τις εξαγωγές. Μειώθηκε από την άλλη η εξαγωγή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ορυκτών από τις χώρες αυτές. Αυτό είναι κάτι το θετικό. Τώρα, κεφάλαιο 6, βιωσιμότητα, σελίδα 62. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μπροστά στην αναπτυξιακή συνεργασία και στην πρόθεση υπεύθυνων πρακτικών ε, δανεισμού. Κεφάλαιο 7. Αντιμετώπιση συστημικών προβλημάτων, σελίδα 66. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προωθήσει την συνοχή πολιτικής για το ζήτημα αυτό και επίσης την ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης ε, των ε, συστημάτων αναπτυξιακής βοήθειας. Στο κεφάλαιο 8 τώρα στη σελίδα 82. Τεχνολογία, επιστήμη, καινοτομία και δημιουργία ικανοτήτων. Βλέπουμε εδώ ότι τα κράτη-μέλη και πάλι είναι στην πρώτη θέση σε ό,τι φορά την παροχή βοήθειας ε, με τη μορφή ε, όχι μόνο χρηματική στήριξη αλλά και υποτροφιών για παράδειγμα για σπουδές. Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η έκθεση που παρουσιάστηκε στο Φόρουμ για την Ανάπτυξη στις 23 ε, Απριλίου στη Νέα Υόρκη είναι θετική η έκθεση. Έχει δείξει πως ε, βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι φορά την επίτευξη των στόχων της Αντίσα Μπέμπα αλλά χρειάζονται φυσικά περισσότερες προσπάθειες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, βλέπουμε ότι στο πίσω μέρος της ε, έκθεσης, από την σελίδα 93 δηλαδή και μετά, βλέπουμε όλους τους εφωτινούς σηματοδότες, βλέπουμε τις ε, δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ένωση. Ε, έχω μια ερώτηση. Η έκθεση αυτή τώρα θα συντάσσεται κάθε χρόνο. Πώς θα συνεχίσετε. Δεν έχουμε λάβει ακόμα αυτή την απόφαση. Σίγουρα του χρόνου δεν θα καταρτιστεί έκθεση, γιατί θα συμπέσει με άλλες εκθέσεις που καταρτίζονται. Δεν έχουμε όμως αποφασίσει ακόμα για το πότε θα καταρτίζεται η έκθεση αυτή. Ναι, βλέπω και εγώ στο πίσω μέρος της έκθεσης ότι όλα βαίνουν ε, καλώς, με εξαίρεση κάποιους τομείς που είναι ανησυχητικοί. Όπως για παράδειγμα ε, αυτό που συμβαίνει με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως ε, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, έκανε μια παρουσίαση σχετικά με το πού βρισκόμαστε, τι πάει καλά, τι όχι, ποια είναι τα προβλήματα. Γιατί έχουμε ένα θέμα με την ενημέρωση. Ορισμένα μέλη της Επιτροπής, μάλιστα, από όσο γνωρίζω, έλαβαν την έκθεση μόλις σήμερα το πρωί και δεν πρόλαβαν να τη μελετήσουν. Επίσης, να σας ρωτήσω τι κάνετε για τη διαφάνεια. πώς ε, ενημερώνετε και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους οργανισμούς για, για τα αποτελέσματα των ερευνών σας. Ναι, να σας απαντήσω. Συναντήθηκα με διάφορους εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων χθες, έτσι ώστε να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα. Όπως είπατε κι εσείς, στην έκθεση στο τέλος της βρίσκεται και αυτό το σύστημα με το φωτεινό σηματοδότη έτσι ώστε να τονίζονται περισσότερο τα επιτεύγματα και τα προβλήματα. Χρειάζεται όμως χρόνος έτσι ώστε οι υπόλοιποι φορείς να αξιολογήσουν τα ευρήματα της έκθεσης και να εξετάσουν τις ε, δράσεις που χρειάζονται. Ωραία. Τότε λοιπόν ε, θα το εκτιμούσαμε εάν ε, ενημερώνατε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα επόμενα βήματα για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Διότι τον Ιούνιο έρχεται και ένα νέο πρόγραμμα, γι' αυτό λοιπόν ε, χρειάζεται να δούμε τι θα κάνουμε ήδη τώρα. Ο Νόρμπερτ, έχεις μια ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Η τεκμηρίωση ήταν εξαιρετική. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί η, πρόεδρο, πρόοδος στην εφαρμογή των ε, στόχων της Αντίσα Μπέμπα. Και είναι επίσης σημαντικό να τηρήσουμε τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει. Με συγχωρείτε, σας διακόπτω. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την ε, διερμηνία. Νομίζω πως ε, έχουν μπλεχτεί τα κανάλια. Τώρα λύθηκε το πρόβλημα. Ναι, ακούτε στα γερμανικά, λέει ο πρόεδρος. Ωραία, Νόρμπερτ, συνέχισε. Ευχαριστώ. Είναι πολύ καλή, λοιπόν, η παρουσίαση. Βλέπουμε τη γενικότερη εικόνα. Βλέπω ότι η εφαρμογή είναι κάτι το οποίο είχε αποφασιστεί για μετά την ε, σύνοδο της Αντίσα Μπέμπα και μπορούμε λοιπόν, θεωρώ, να συνεχίσουμε να καταρτίζουμε εκθέσεις κάθε χρόνο. Ίσως όχι μία νέα έκθεση, αλλά διάφορες ε, εκθέσεις παρακολούθησης για να δούμε τι γίνεται στη συνέχεια. Πολύ σημαντικό για μένα είναι να συμπεριληφθεί η ανάπτυξη στην ημερήσια διάταξη στα κράτη-μέλη. Όταν συζητούσαμε το θέμα της συνένεσης για την ανάπτυξη, κάποια κράτη-μέλη είχαν παρουσιάσει ε, προβλήματα στην επίτευξη του στόχου του 0,7%. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε την ανάπτυξη στα διάφορα κρατημέλη και όχι να αρκεστούμε στο να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ε, αναπτυξιακής βοήθειας. Να δούμε τι γίνεται και στο κάθε ένα από τα κρατημέλη. Και συμπεριλαμβάνεται και η δική μου χώρα σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό θεωρώ να δούμε ποια μέσα έχουμε στη διάθεσή μας έτσι ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Δεν είναι καλό σημάδι ότι αυτές οι χώρες ε, παρουσιάζουν προβλήματα. Αυτό δείχνει έλλειψη στήριξης από δική μας πλευρά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Μαρία Χόιμπουχ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την... Με ακούτε? Τώρα με ακούτε. Και εγώ θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για αυτήν την ε, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και περιεκτική έκθεση. Νομίζω πως εξετάσατε με αρκετή λεπτομέρεια το τι γίνεται στα κράτη-μέλη, όμως ο Νόρμπερτ ε, κατονόμασε ορισμένα πράγματα, ορισμένα προβλήματα και πρέπει νομίζω να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες παρατήρησα και εγώ πως ε, είναι ένα μελανό σημείο και όπως είπε και η Λίντα και ο Νόρμπερτ, είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε, να δούμε πού είναι τα προβλήματα, να δούμε γιατί δεν έχουν καταφέρει κάποια κράτη-μέλη να επιτύχουν το στόχο του 0,7%. Να αναφερθώ λίγο και σε ένα άλλο κεφάλαιο για τη βιοπικιλότητα που αναφέρεται στο κεφάλαιο 4,5. Εδώ, τι συμβαίνει με την χρηματοδότηση για τη βιοπικιλότητα των οικοσυστημάτων. Αναφέρονται υποχρεώσεις για τα κράτη-μέλη που προκύπτουν από την ε, διάσκεψη για τη βιοπικιλότητα του 2010. Αναφέρεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί, όμως οι στόχοι ε, χρηματοδότησης για το 2020 είναι ελλειπής. Εδώ βλέπω πως υπάρχουν κάποιες ε, συμφωνίες. Γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρώ πως ε, πρέπει να καλυφθούν αυτά τα κενά και σίγουρα η χρηματοδότηση της βιοπικιλότητας είναι κάτι πολύ δύσκολο, διότι οι ιδιώτες επενδυτές ε, δεν έχουν το ενδιαφέρον που χρειάζεται. Και η χρηματοδότηση λοιπόν επιβαρύνει το δημόσιο τομέα. Πώς θα λύσουμε όμως αυτό το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση για τη βιοπικιλότητα και πρέπει να ε, προσελκύσουμε και ιδιωτικό κεφάλαιο. Ε, μετά βλέπω ιδιαίτερα αισιόδοξη στάση για την ε, χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Βλέπω λοιπόν ότι η έκθεση τα παρουσιάζει πολύ θετικά τα πράγματα. Και θέλω να ρωτήσω, εσείς πώς καταλήξατε σε αυτά τα συμπεράσματα. Πώς θεωρείτε πως το επενδυτικό σχέδιο της Ευρώπης θα καταφέρει να προσελκύσει ε, τον ιδιωτικό τομέα ε, έτσι ώστε να διαθέσει πόρους για την βιοπικιλότητα αφού προηγουμένως στην έκθεση μας λέτε πως ε, υπάρχουν ελλείψεις σε αυτό το τομέα. Πώς θα το καταφέρετε αυτό και ποια είναι τα κεφάλαια που αναμένεται να διατεθούν για την βιοπικιλότητα. θα καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τους στόχους χρηματοδότησης ε, για το 2020. Εδώ δεν βλέπω ε, να υπάρχει γενικότερα πολύ... Δεν, δεν βλέπω να υπάρχουν λεπτομέρειες. Και αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και επίσης η χρηματοδότηση προς τους ε, γεωργούς, προς τη γεωργία. Βλέπω κάποια προβλήματα και θα ήθελα λοιπόν να σας ε, υπενθυμίσω ότι δεν έχουν δοθεί οι απαντήσεις που έχουμε ζητήσει. Σας ευχαριστώ. Αν δείτε τα παρατήματα και από την ε, σελίδα 170 και μετά υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε κράτος μέλος, τις τάσεις, κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Από τη σελίδα 170 και μετά στα παρατήματα βλέπουμε την, ε, το παράδειγμα της Γερμανίας. Όπως είπε ο Νόρμπερτ, θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Μπόγκναν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τη σημασία του, ε, της Ευρωπαϊκής Συνένεσης για την ανάπτυξη. Μπορούμε να πούμε ότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 0,7% είναι σημαντικός, αλλά πρέπει να δούμε πώς κατανέμονται οι προσπάθειες σε κάθε κράτος μέλος. Πολύ σημαντικό να κάνουμε διάλογο με τα κράτη-μέλη, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα και σε συνεργασία με συναδέλφους από την Επιτροπή Προϋπολογισμού ε, γίνονται συζητήσεις για το τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Λόρα. Σε ευχαριστώ. Εμεί μέσα στο ίδιο με μια από το 2017 είχαμε και πάλι μια συνένεση για την ευρωπαϊκή πολιτική ανάπτυξη για να προχωρήσουμε για το 0,7 αλλά σύμφωνα με το DAC του περασμένου μήνα το 2017 η ε, ενίσχυση ανέβηκε στο 6,7% σχέση με το 16 και έχουμε κάποιες χώρες που το πέτυχαν το 0,7 αλλά θα πρέπει να δούμε αν θα κάνει φιλοπορίας η Κομισιόν που να είναι ρεαλιστικό για αυτές τις ε, υποσχέσεις που έχουμε δώσει. Το έχεις δει στο κοινοβούλιο πανελλημένα. και να δούμε πώς θα τα μπαλώσει η Κομισιόν όσον αφορά ε, το έλλειμμα ούτως επίν των πόρων που θα προγύψει από το Brexit ή πρόεδρος. Θα συζητήσουμε το απόγευμα, θα έχουμε κάποιους ειδικού που θα έρθουν για να δούμε τι γίνεται σε επιπτώσεις του Brexit. Έχει διάλογος το λόγο. Οπότε έχετε εσείς το λόγο. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Βασικό σημείο σε αυτή την έκθεση είναι το τι κάνει όλοι μαζί η Ένωση, τι κάνει το κάθε κράτος μέλος και πού βρίσκεται το καθένα σχέση με τις ε, υποχρεώσεις. Τώρα όσον αφορά την αύξηση της νευρωσιακής βοήθειας το 2017 και ε, τη, τιμήωση, η βασική λόγη είναι η εξής. Πρώτα-πρώτα έχουμε αυτά τα επιλέξιμα έξοδα για τους πρόσφυγες. αυτή η δαπάνη παραμένει. Μια που συνεχίζεται να υπάρχει το πρόβλημα και θα συνεχιστεί για τα επόμενα δύο-τρία χρόνια. Επίσης κάποια κρατημέλη ακύρωσαν κάποιες κινήσεις του 16, οπότε αυξήθηκε το ότι έγινε τη χρονιά, δεν επανέλθει το 17. Επίσης, από την ΕΤΕ έχουμε κάποια δάνεια επί τη βάση ταμιακών ροών και θεωρήθηκαν ε, αυτές οι ροές ως αρνητικά ODA. Οπότε τώρα το 2017 είχαμε αύξηση αυτών των ροών, οπότε αυτομάτως μειώθηκε η αμυσιακή βοήθεια των θεσμικών οργάνων. Να γιατί έχουμε συνολική μείωση πάντως ακόμη ανησυχούμε που έγινε το 17 αυτή η μείωση της αντίστοιχη βοήθειας και στις 22 Μαΐου το Συμβούλιο ελπίζουμε να εγκρίνει στα συμπεράσματα το ότι ζήτησε από την Κομισιό να ξεκινήσει κάποιες πρωτοβουλίες κάποιες προτάσεις τόσο ώστε οι υποσχέσεις για την εμπιστική βοήθεια να τηρηθούν αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει Πάντως τα πράγματα επίγουν, πιέζουν και θα πρέπει επομένως να λάβουμε υπόψη ότι αυτή η ένευση έχει βοηθεί αφορά τις λιγότερο αντιγμένες χώρες. Αυτά για το σύμβολο Και θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι ειδική κατηγορία οι λιγότερο αντιγμένες χώρες και δεν είναι όλες ευάλωτες. Και ούτε όλες οι ευάλωτες είναι λιγότερο αντιγμένες αλλά θα πρέπει να τα αναλύσουμε καλύτερα. Πάντως ένας βασικός χώρος, βασικός λόγος συγγνώμη, είναι το, του γιατί κόλλησε η βοήθεια προς αυτά τα LDC είναι ότι πρόσφατα πάρα πολύ βοήθεια πήγε σε κάποιες σε ευάλωτες χώρες που δεν είναι λιγότερο από τις χώρες και έχουμε πάρα πολλούς πρόσφυγες σε σχέση με, με το Συριακό και ευθύγησαν κάποιε χώρε που είναι λιγοτομικές χώρε, αλλά δεν είναι αναγκαστικά όλε ευάλωτε. Ε, αυτό εξηγεί το γιατί τα λιγοτομικές χώρε δεν πήραν αρκετά, αρκετού πόρου. Τέλο πάντων αυτό δεν είναι για να μα καθησυχάσει αλλά έτσι έχει η κατάσταση. Οπότε για να δούμε τώρα τι γίνεται με τη διμερή βοήθεια, τι δομή έχει. να το αναλύσουμε και κατόπιν να δούμε τι πρόταση θα διατυπώσουμε, τόσο να βελτιωθεί η κατάσταση για την βοήθεια προς τις χώρες εκείνες. Τώρα σου με τη βιοποικιλότητα δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να σας πω κατά λεπτό στην απάντηση γιατί δεν είμαι ειδικό. Αλλά ούτε για το EIP ούτε για την βιοποικιλότητα. Αλλά δεν ενδιαφέρει ιδιωτέρως ο ιδιωτικός τομέας για την βιοποικιλότητα. Και είναι από του στόχου τη ε, EIP αυτό, το να κατευθύνει προ εκεί ο ιδιωτικό τομέα. Και με μεικτή χρηματοδότηση ελπίζουμε ότι ο ιδιωτικό τομέα θα συμμετάσχει εκεί που δεν θα το έκανε και για τη βιοποικιλότητα. Τα λέμε στην έκθεση και ελπίζουμε ότι αυτό θα βγει σε βελτίωση. Θα το πω στους συναδέλφους που ασχολούνται με το EIP. Και για την ερώτησή σας τότε ε, θες το καλή εβδομάδα να σας απαντήσουν. Να δούμε πώς θα υπάρχει χρηματοδότηση. Πολύ σημαντικό αυτό. Ε, κάτι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε πόσο αποτελεσματική θα είναι όμως το μέλλον για αυτές τις χρηματοοικονομικέ ζωές. Πολύ σημαντικό. Για τα επόμενα χρόνια και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να μας ενημερώνει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και θα παρακολουθούμε για να δούμε πού υπάρχουν ε, προβλήματα σχέση με τις λιγότερο αντιμονές χώρες Είπαμε ότι να συζητηθεί το θέμα της ε, Ουγγάντα και υπάρχει θέμα με, έργα, προγράμματα, σχέδια και εκεί θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το μεταναστευτικό. Συνεχίζει και τρέχει το σχετικό πρόγραμμα. Ευχαριστούμε την Επιτροπή που μας ε, ενημέρωσε. Κοιτάξτε επομένως το ντοσιέ, τα έγγραφα, να δείτε τι κάνει η δική σας χώρα και σας ευχαριστούμε πολύ. Can we thank the guest speaker? Thank you. Thank you very much. Okay, we now move on. We've got a lot of important issues this morning. Συναδελφοί, έχουμε πολλά σημαντικά θέματα. Το επόμενο είναι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα καλέσουμε τους επιτρόπους σήμερα και αύριο για να συζητήσουμε τις νέες προτάσεις. Σήμερα όμως θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων με την Concord για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς και με την πολυμερή πλατφόρμα για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Πού κάθεστε? So, we Λοιπόν, συνάδελφοι, όλοι είδαμε στην Ολομέλεια τον πρόεδρο Γιούνκερ να παρουσιάζει την πρόταση για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνδυάζει διάφορα χρηματοδοτικά μέσα σε ένα το οποίο ονομάζεται μέσω ε, για τη γειτονία, την ανάπτυξη και τη διεθνή συνεργασία. Η πρόταση αυτή λοιπόν συνδυάζει όλα αυτά και τα εισαγάγει στον προϋπολογισμό. Εμείς ε, έχουμε ως στόχο η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη να παραμείνει κύριο σημείο στο νέο αυτό πρόγραμμα, εάν δηλαδή το Κοινοβούλιο δεχτεί αυτή την ενοποίηση των ε, μέσων. Κάποιοι από εμάς ε, πριν από δύο εβδομάδες παραβρέθησαν στη συνεδρίαση με την ε, Concord. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από την Κομισιόν. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πολύ που καλωσορίζω και σήμερα την εκπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών, έτσι ώστε να συζητήσουμε τις προτάσεις της Επιτροπής. Η Καταρίνα Λεμάνσκα, εκπρόσωπος λοιπόν της Concord, ο Ραφαήλ Βέιλαντ από την ε, Νάμπου ε, Βρυξέλλες, εν περιβαλλοντική οργάνωση και είναι και εισηγητής για την έκθεση σχετικά με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα μπορούσατε ίσως να μας πείτε δύο λόγια για το τι κάνετε. Θα δώσω λοιπόν το λόγο σε εσά ε, για να μας παρουσιάσετε τις εντυπώσεις σας από τη νέα πρόταση της Επιτροπής. Ποια είναι τα καλά και τα όχι τόσο καλά σημεία. κυρία Λεμάνσκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να έρθω και να συζητήσουμε το την πρόταση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και την εξωτερική δράση. Ονομάζομαι Κατερίνα Λεμάνσκα, εκ μέρου ε, τη ε, Concord. Εργάζομαι επίση και στην Global Health Advocates. Όπω γνωρίζετε, η Concord είναι συνομοσπονδία οργανώσεων ε, για την ανάπτυξη. Σε εμά βρίσκονται 28 εθνικές πλατφόρμες και 21 διεθνή δίκτυα τα οποία αποτελούνται από 2.600 ε, οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν ε, σήμερα είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα του συλλογικού μας ε, έργου. Το 2015 λοιπόν μας έκανε όλους περήφανους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε έμφαση στα δίδυμα, όπως τα είπε ο Μπάνκι Μουν, σχέδια για την διαδικασία μεταμόρφωσης. Γνωρίζαμε ότι η διαδικασία εφαρμογής θα ήταν κάτι το δύσκολο, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται και ανάληψη δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Φυσικά δεν γίνεται να μην επιτευχθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης διότι διαφορετικά ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος θα είναι τεράστιος. Ελπίζουμε λοιπόν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και η Συμφωνία του Παρισιού να αποτελέσουν ε, τα πρότυπα για την εφαρμογή των στόχων αυτών. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζουμε την πρόταση της Επιτροπής να ε, αυξηθεί η χρηματοδότηση κατά 30% μάλιστα ε, δεδομένων των μειωμένων πόρων ως αποτέλεσμα του Brexit. Βέβαια, θα θέλαμε να υπάρχουν και διασφαλίσεις ότι θα διατηρηθούν τα ίδια επίπεδα χρηματοδότησης και στο μέλλον, στο επόμενο κεφάλαιο. Η δομή λοιπόν ε, του πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι έχει ως εξής. Το 2011 στην πρόταση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παρουσίασε ένα σιαφή διαχωρισμό των πόρων και ανέλαβε τη δέσμευση να διαθέτει το 0,7% του ΑΝΕΠ για αναπτυξιακή βοήθεια. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι την εποχή εκείνη η υιοθέτηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης θεωρήθηκε ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα πρέπει να αυξηθούν οι πόροι για εξωτερική δράση. Όχι μόνο να αυξηθεί η συνεισφορά ε, στο 0,7% του ΑΕΠ. Τα κράτη-μέλη πρέπει τα ίδια να ε, τηρούν τις ε, υποσχέσεις τους. Δεδομένου μάλιστα, δεδομένης μάλιστα της ε, κατάστασης αυξημένης ε, πίεσης λόγω του μεταναστευτικού, του προσφυγικού κτλ. Χρειάζεται λοιπόν ε, αναπροσαρμογή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης έτσι ώστε να ανταποκρίνεται ε, στις ε, νέες απαιτήσεις. Ανησυχούμε όμως ότι αυτή η αναπροσαρμογή θα απομακρυνθεί από τους μακροπρόθεσμους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Η πρόταση λοιπόν είναι να συγχωνευτούν 12 μέσα τα οποία υλοποιούν ε, ένα εύρος ε, πολιτικών. Για παράδειγμα, αναπτυξιακή πολιτική, πολιτική γειτονία, ανθρώπινα δικαιώματα, ειρηνευτικές ε, διδικασίες και αυτό θεωρούμε πως θα αποδυναμώσει τους επιμέρους στόχους και θα κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια, Πρώτον, η νέα δομή έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί καλύτερα τις προτεραιότητες της Ένωσης. Φυσικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να, να ενεργήσει αυτόνομα για, τα, για τους εδικούς της ε, στόχους. Αυτό που δεν βλέπουμε στην πρόταση είναι σαφείς δεσμεύσεις για τη διαφύλαξη της ακυριότητας των ε, κυριότερων ε, στόχων η μετανάστευση έχει γίνει προτεραιότητα και αυτό νομίζω πως ε, δείχνει ξεκάθαρα την αλλαγή των προτεραιοτήτων. Πρέπει να δούμε την ανάπτυξη μέσω της μετανάστευσης και η ιεράρχηση της μετανάστευσης δείχνει τη να αλλαγεί στη συγκυρία. Εμείς θα περιμέναμε την ισότητα των φύλων και την προστασία των πολιτών να είναι στην κορυφή. Απαλυφή της φτώχεια, να ανέβει πιο πάνω στον κατάλογο προτεραιοτήτων, αύξηση των δαπανών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Βέβαια, δεν πιστεύουμε κατά ανάγκη ότι υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στους ε, στόχους της Ένωσης και ε, σας παρακαλώ να μιλάτε πιο αργά, λέει η Πρόεδρος, για να μπορεί να γίνει και διερμηνία. Συνεχίζω λοιπόν. Υπάρχει κάποια συμφωνία και κάποιες εντάσεις. Δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε τονίσει τα προβλήματα αυτά. Αν δούμε την ενδιάμεση αναθεώρηση του EDF θα παρατηρήσουμε ότι αυτές ε, οι εντάσεις είναι κάτι το φυσιολογικό, όμως πρέπει να αντιμετωπιστούν και πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητά μας αυτό. Στην παρούσα πρόταση λοιπόν δεν βλέπουμε να έχει ληφθεί υπόψη η σύσταση αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλά εκρεμή ζητήματα, για παράδειγμα διακυβέρνηση των, ε, και διαχείριση των μέσων αυτών. Δεν γνωρίζουμε από πού θα προέρχεται η πολιτική καθοδήγηση. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος θα διαμεσολαβεί ανάμεσα στα συγκρόμενα συμφέροντα. Δεν γνωρίζουμε από πού θα προκύψουν οι πόροι και δεν γνωρίζουμε ούτε και το ρόλο του Κοινοβουλίου. Η συμβατότητα επίσης είναι ένα φλέγον θέμα σε σχέση με την προσαρμογή ε, του μέσου στο μέλλον και στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτιμά την ευελιξία παρά την ε, ικανότητα προσαρμογής. Ωστόσο, δεν αναφέρει πώς θα γίνει αυτό και πώς θα αποφευχθεί να υπονομεύσουν οι νέες προτιμόμενες δράσεις ε, τους αναπτυξιακούς στόχους. Έπειτα, είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να δημιουργήσει ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκριση σε τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχει κάποια πρόταση για μηχανισμό ευελιξία στα πλαίσια του πολιτούς δημοσιονομικού πλαίσιου. Υπάρχει λοιπόν αρκετή ευελιξία, υπάρχουν αρκετά διάθετα ποσά. Δεν ξέρουμε λοιπόν πώς ε, θα γίνει η διαχείριση των πόρων αυτών. Παρατηρούμε μία εσωστρέφεια στην ε, διαχείριση των πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα εσωστρέφεια εκεί που παλαιότερα υπήρχαν ε, στόχοι προτεραιότητας. Θεωρούμε πως αυτό είναι ενδεικτικό του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει το ενδιαφέρον της για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων και εστιάζει περισσότερο στους βράχυπρόθεσμους στόχους. Επίσης, ε, είναι ενδεικτικό ότι οι πιο ευάλωτες ε, περιοχές θα μείνουν εκτός και θα δοθεί έμφαση στις ε, γεωπολιτικά σημαντικές περιοχές. Αυτό θεωρώ πως πρέπει να επισημανθεί, ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι πιστεύουμε ότι τόσο για εμάς όσο και για εσάς θα είναι αρκετά δύσκολο εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν οι στόχοι εάν ε, το εύρος των δραστηριοτήτων ε, είναι μεγάλο, εάν καλύπτονται πολλές περιοχές με τους ίδιους στόχους. Γι' αυτό δεν πιστεύουμε ότι το μέσο αυτό θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσει επαρκώς ε, τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Σίγουρα μπορεί να επιτευχθεί απλούστευση, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ε, υλοποίηση των στόχων και των διεθνών δεσμεύσεων. Τώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Τα επόμενα βήματα θεωρούμε πως χρειάζεται βιώσιμη πολιτική διαχείριση και για μας ως ε, Concord είναι πολύ σημαντική η δημιουργία ενός χρηματοδοτικού μέσου το οποίο θα καλύπτεται 100% από πόρους και θα στοχεύει στην απαλληλή της στόχης και στην ε, επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης πρέπει να μην χάσουμε την έμφαση στην ε, πολιτική γειτονία και τα διάφορα σχετικά μέσα. Επίσης, θα επιμείνουμε στην ε, κάλυψη του 90% των ε, στόχων του κεφαλαίου αυτού Οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη, το κλίμα και η ισότητα πρέπει να συμπεριληφθούν σε όλες ε, τις ε, πολιτικές Ευρωπαϊκή Ένωσης. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα ε, σημεία προόδου για τους στόχους αυτούς. Και τέλος, η κοινωνία των πολιτών πρέπει να έχει τα δικά της ε, προγράμματα και τους δικούς της ε, πόρους καταναμημένους ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν ε, από περιοχή σε περιοχή. Θα ήθελα τέλος να σας πω ότι η δική μας θέση και η δική μας πρόταση καλύπτει πολλούς από αυτούς τους τομείς, αλλά να κλείσω λέγοντας ότι πρέπει να διασφαλίσουμε πως θα ακούγονται οι φωνές οι δικές μας και οι δικές σας. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, οι ΜΚΟ δεν ε, είναι ευχαριστημένε με αυτή την ενοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων, όπω ε, είπε και η Κονκόρντ. Ράφελ, ο, έχει το λόγο. Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Σήμερα ε, συζητάτε για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της επιπτώσεις για την συνεργασία. Προσωπικά δεν είμαι ειδικό ε, σε θέματα ανάπτυξης, αλλά θα ήθελα να πω κάποια ε, πράγματα σχετικά με αυτό. Λέγομαι Ράφαελ Βέλαμαν, εργάζομαι για τη Γερμανική Περιβαλλοντική Οργάνωση ΝΑΜΠΟΥ, που ανήκει στην BirdLife Europe. Ήμουν εισηγητής της έκθεσης για το MFF της ε, πολυμερούς ε, πλατφόρμας για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ε, την οποία παραδώσαμε στον Αντιπρόεδρο Τίμερμαντς. Και η έκθεση αυτή δημοσιεύτηκε στο site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αυτή την έκθεση και με άλλες εκθέσεις, άλλες οργανώσεις, στα πλαίσια της Concord, παρακολούθησα τις συζητήσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω πιο γενικά για την ε, υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό που θα πω είναι μεν γενικά, αλλά είναι σημαντικά. Πιστεύουμε ότι δεν αρκεί να ε, εστιάσουμε μόνο στις γραμμές χρηματοδότησης που αφορούν τη συνεργασία για την ανάπτυξη. όλες οι δαπάνες στα πλαίσια του ε, MFF πρέπει να είναι βιώσιμες. Για ποιο λόγο, γιατί οι δαπάνες Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν επιπτώσεις και ε, πέρα από τη σύνορα της Ένωσης. Το, σύμφωνα με το σημερινό MFF, 40% των δαπανών πάνε στην κοινή γεωργική πολιτική. Η κοινή γεωργική πολιτική εστιάζει στις άμεσες ενισχύσεις και έτσι αποτυχάνει να επιτύχει τους στόχους της σε οικονομικό, κοινωνικό και οικολογικό επίπεδο. Τον Μάρτιο η Euroactive δημοσίευσε μια μελέτη δείχνοντας ότι η παραγωγή ε, γάλακτος σε σκόνη ε, στην, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει ε, αρνητικά την παραγωγή στην Αφρική. το σημερινό, το εφιστάμενο πολιτές δυναμικό, δημοσιονομικό πλαίσιο δεν προβλέπει επαρκή ανάλυση της κατανομής των δαπανών. Και ε, καταλήγουμε να χρηματοδοτούμε πολιτικές που έχουν αρνητικές ε, επιβλαβείς επιπτώσεις για το κλίμα. Ε, αυτό το βλέπουμε και ε, με δράσεις στα πλαίσια του σχεδίου Horizon και ε, των πανευρωπαϊκών δικτύων για τις μεταφορές και την ενέργεια. και όμως οι περισσότερο ευάλωτες περιοχές στην κλιματική αλλαγή βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό αυτό ε, συστήνουμε την ε, ένταξη διαφόρων οριζόντιων ε, μέσων για την προσαρμογή του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και συγκεκριμένα συστήνουμε. Χτες ο ε, Επίτροπος δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει άλλο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο πριν την ολοκλήρωση του θεματολογίου του 2030. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να δράσουμε. Το σημερινό πλαίσιο λύγει τουλάχιστον μέχρι το 2027. Οι υλοποίηση των δράσεων του θεματολογίου ε, προβλέπονται μέχρι το 2030. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν χρειαζόμαστε νέες γραμμές χρηματοδότησης, ούτε αύξηση των δαπανών. Πρέπει να ε, σταματήσουμε την, ε, τις αντιφατικές ε, δράσεις. Πρέπει λοιπόν να εντάξουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, δράσεις που χρηματοδοτούμε, προκειμένου να υπάρχει συνεκτικότητα. Τρίτη σύσταση, θα έπρεπε να υπάρξει ένας έλεγχος της βιωσιμότητας των δράσεων η ομάδα εμπειρογνωμόνων, εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου έχει προτείνει τη χρήση της αρχής ε, ε, της βιωσιμότητας, το Think Sustainability First, για οποιαδήποτε δράση ε, χρηματοδοτείται. Είναι σημαντικό λοιπόν και οι αξιολογήσεις επιπτώσεων να διασφαλίζουν την βιωσιμότητα των δράσεων. Επίσης, ε, πρέπει να ε, εστιάσουμε σε χρηματοδοτήσεις και δαπάνες που δεν είναι πλέον ε, βιώσιμες. Αυτό ισχύει κυρίως στο τομέα της γεωργίας, της βιοποικιλότητας και για τη χρηματοδότηση των υποδομών. Η έκθεση προτείνει και άλλα χρηματοδοτικά μέσα, αλλά θα ήθελα να εστιάσω στο εξής θα πρέπει να μεταβούμε σε μια προσέγγιση που είναι πιο διαφανής και βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δημοσίευσε την ε, εξέταση των δαπανών ε, πριν παρουσιάσει την ε, πρόταση του Επιτρόπου Έτιγκερ Μπορεί κάποιοι από εσά να πιστεύουν ότι το πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είναι τόσο σημαντικό. Είναι, πιστεύω ότι είναι θέμα των συναδέλφων σα από την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Όμως, όπω είπε ο πρόεδρο Γιούγκερ πριν από λίγο καιρό, δεν πρόκειται μόνο για ε, εργαλείο ε, χρηματοδότησης. Ε, το MFF χρησιμοποιείται και για την επίτευξη πολιτικών στόχων. Γι' αυτό, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, ε, σας, προτείνω να μην δεχτείτε ως έχει την πρόταση της Κομισιόν για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί έτσι όπως προτείνεται και συνεχίζει να εστιάζει στις άμεσες ενισχύσεις οι οποίες είναι αναμοτελεσματικές και μη βιώσιμες. Και κάτι τέτοιο δεν θα είναι αρκετό για να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού και δεν υπάρχει καμία συνεκτικότητα και ε, καμία προσαρμογή στους στόχους βιώσιμης ε, ανάπτυξης. Αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη της Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλει να κερδίσει την ε, εμπιστοσύνη των πολιτών. Στο χέρι των κρατών μελών είναι να, τώρα να συζητήσουν για το ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά έχει ρόλο να παίξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ωραία. Και έτσι μας αναλύσατε τα του πολιτού του δημοσιονομικού πλαισίου όσον αφορά την ανάπτυξη και είδαμε τι γίνεται να υπάρχει βιωσιμότητα. Πολύ ενδιαφέρον. Άδελφε, έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα του δώσουμε το λόγο. Αλλά πρώτα-πρώτα οι συνάδελφοι. Μαρία, πρώτη. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Φορέστε τα ακουστικά σας, παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις παρουσιάσεις σας και ευχαριστώ πολύ ιδιαίτερα την κυρία Λεμάντσκα διότι πραγματικά είπατε αυτά που εμείς θεωρούμε σημαντικά ως Επιτροπή Ανάπτυξης και επισημάνατε και τα ίδια προβλήματα που έχουμε επισημάνει και εμείς. Η ευελιξία, όπως παρατηρήσατε κι εσείς, έχει ε, προβλήματα. Υπάρχουν ασάφειες, δεν γνωρίζουμε ποιος θα ελέγχει τι, ε, ποιοι διάβλοι θα χρησιμοποιηθούν στην ε, διαχείριση, ποιοι θα είναι υπεύθυνοι. Αυτό το 20% των πόρων, όπως είδαμε, θα διατίθεται για την ευελιξία, αλλά δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει, πώς ε, θα ε, διαθέσουμε κονδύλια για την καταπολέμηση της ε, φτώχειας. Κύριε Βάιλαντ, αναφέρατε πάρα πολύ σημαντικά θέματα, για παράδειγμα την ε, γεωργική πολιτική, κάτι που εμείς ε, θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Να είστε λοιπόν σίγουρος ότι η Επιτροπή Ανάπτυξης και η Επιτροπή Γεωργίας παίρνουν το θέμα αυτό πάρα πολύ στα σοβαρά. Ε, να μην ξεχάσω και την Επιτροπή Προϋπολογισμού, η οποία θα πρέπει να εγκρίνει τις νέες γραμμές του προϋπολογισμού. Ε, εκτός από το Συμβούλιο και εμείς ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή με το θέμα. Τώρα, η γεωργία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη βιωσιμότητα στην Ευρώπη και παγκοσμίω βλέπουμε ότι αν θέλουμε να επιτύχουμε οτιδήποτε υπέρ της βιοπικιλότητας, ε, υπέρ του περιβάλλοντος, των υδάτων, της ποιότητας των υδάτων κτλ. πρέπει να το δούμε αυτό σε συνδυασμό με την ε, γεωργία. Επίσης, σε ό,τι αφορά τι άμεσες ενισχύσει, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις για τις άμεσες ενισχύσεις. Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για τη γεωργία δεν θα, έπρεπε, δεν ε, θα έπρεπε να υπάρχει αυτό, διότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε τους ε, στόχους μας διαφορετικά. Βλέπουμε ήδη από τις ε, γενικότερες γραμμές που, προς τα η κατάσταση, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει η ίδια τάση και για την αναπτυξιακή συνεργασία. Στηρίζουμε διάφορα γεωργικά ε, έργα και προγράμματα, όμως ας ε, το δούμε με περισσότερη προσοχή και ας δούμε πώς από αυτά τα προγράμματα αφορούν την βιώσιμη γεωργία. Θα δείτε ότι είναι ελάχιστα. Η συνάδελφοί μου που ασχολούνται με την γεωργία θα σας το επιβεβαιώσουν ότι η βιολογική γεωργία ε, έχει να κάνει με την ε, κυκλική οικονομία, την κυκλική γεωργία, την ε, βιοπικιλότητα, τη βιωσιμότητα, αλλά υπάρχουν και άλλες διαστάσεις, κοινωνική διάσταση. Ο άνθρωπος βρίσκεται, όπως και το περιβάλλον, στο επίκεντρο. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, χρειάζεται αύξηση σταδιακά της ε, βιολογικής γεωργίας και αυτό πιστεύω πως είναι κάτι που ε, αγνοούμε κάπως ε, στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή σε αυτό. Πρέπει να κοιτάξουμε τι ακριβώς ζητάνε στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και να μην ξεχνάμε το πώς αυτοί συνδέονται με την βιολογική γεωργία. Ευχαριστώ πολύ. Θα συζητήσουμε με τον Επίτροπο Μίμητσα αύριο το πρωί για τα θέματα αυτά. Ο Σαλ Γκέρεντς στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τις δύο παρουσιάσεις και οι οποίες θα, ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις ε, σχετικά με όσα υπόθηκαν. Επιμείνατε ε, την ε, ε, προτεραιότητα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Πολύ καλά, αλλά δεν πιστεύετε ότι αυτή η προτεραιότητα έχει ως στόχο να διορθωθούν τα λάθη του παρελθόντος. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεωρεί ότι η μετανάστευση είναι προτεραιότητα και, και σε αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις και όχι τις αιτίες του προβλήματος. Θεωρούμε ή περιμένουμε ότι το επόμενο ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα είναι ένα εργαλείο διόρθωσης των λαθών του παρελθόντων. εγώ πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Να ορίσουμε τις προτεραιότητές μας, για να είμαστε ξεκάθαροι, υπάρχουν κονδύλια για την ανάπτυξη, και όλα τα τμήματα που δεν έχουν επαρκή κονδύλια θα προσπαθήσουν να τα αξιοποιήσουν. Η, η πρόκληση λοιπόν θα είναι η ε, κατανομή των κονδυλίων που είχαν αρχικά ε, προβλεφτεί για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Είναι επικίνδυνο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και μετά το Brexit θα παραμείνει πολύ σημαντικός παράγοντας στην, πολιτική, στην αναπτυξιακή πολιτική. Ξέρουμε επίσης ότι θα είναι πολύ δύσκολο να οριοθετήσουμε τις θέσεις μας ε, σε έναν κόσμο όπου ε, ο πρόεδρος των είπα. Ε, απαρνείται τα όσα έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα. Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει. Και αυτή η απάντηση πρέπει να είναι φανερή στο επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν μπορεί να είναι πλήρης αν η Ευρωπαϊκή Ένωση βασιστεί αποκλειστικά στον προϋπολογισμό και το 80% της εξωτερικής ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζεται ε, από τα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να προσθεθεί μια πολιτική διάσταση σε αυτή την προσέγγιση για να συντονίσουμε τις προσπάθειες μας. Είναι απολύτως απαραίτητη η συνεργασία, προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας η ε, ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης γύρει πολλά ερωτήματα. Και όσο το σκέφτομαι, τόσο λιγότερο δογματικός είμαι σε ό,τι αφορά το θέμα. Η εγγραφή αυτών των θεμάτων στον προϋπολογισμό δεν είναι ε, δόγμα, γιατί το σημαντικό είναι να πετύχουμε το αποτέλεσμα. Ε, αν στο τέλος έχουμε λιγότερα κονδύλια, με τα ε, κονδύλια για την ε, ανάπτυξη, για τη συνεργασία για την ανάπτυξη και το ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Αν το αποτέλεσμα λοιπόν είναι η μείωση των κονδυλίων, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Υπάρχουν πολλές ασάφιες, πολλές επικίνδυνες ζώνες και σε ό,τι αφορά την ευελιξία. Ε, πρέπει να δούμε ποια θα είναι η άποψη της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Όπως και να ήθελα να επισημάνω κάποια θέματα για να εκφράσω και τις ανησυχίες μας και να προσθέσω και κάτι άλλο. Το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα θέσει ε, σε αντίθεση όλα τα τμήματα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ε, ανάπτυξη, κοινή γεωργική πολιτική, για παράδειγμα. Και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ε, συζητήσουμε αυτά τα θέματα, να γύρουμε τα απαραίτητα ζητήματα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη την κοινή γεωργική πολιτική, η οποία θα επηρεαστεί και αυτή από ε, αυτά που κάνει ο Τραμπ. Θα υπάρξουν επιπτώσεις και στην εμπορική πολιτική. Θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις ε, και ε, στα πλαίσια των συζητήσεων για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ήθελα λοιπόν να σας προειδοποιήσω ε, δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά αφελείς σε αυτές τις συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει όντως να γίνει συζήτηση και όταν έρθουν οι επίτροποι θα έχουμε αυτή την ευκαιρία. Ιγνάσιο Κορεάλ. Ευχαριστώ, Συμφωνώ. Καταρχήν με όλες τις επιφυλάξεις του Σαλ Γκόρεντς. Πάντως σας ευχαριστούμε για αυτά που μας είπατε και ιδίω εκεί που αναφέρεστε σε αυτό το ε, μοναδικό μέσο χρηματοδότησης για την ε, ευελιξία που δίνει το ότι είναι μοναδικό αυτό το μέσο γιατί ε, έτσι αποφεύγουμε την αναβολή, την μετάθεση της χρήσης των παλιωτέρων μέσων χρηματοδότησης και έτσι τώρα προχωρούμε προς την προτεραιότητα που έχουμε τάξει, δηλαδή τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Οπότε έτσι θα πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε τα μέσα αναπτυξιακής πολιτικής, να ακολουθήσουμε την λογική της θέσπισής τους. Πολύ συχνά έχουμε ε, κάποιο είδου θεή ζώνη στην οποία δίνεται βέβαια η προτεραιότητα στο μεταναστευτικό αλλά υπάρχουν κάποιες ασάφειες εμείς εδώ είμαστε το αντιπροσωπευτικό θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπότε θα πρέπει να διαχειριζόμαστε με διαφάνεια τη χρηματοδότηση τους πόρους που υπάρχουν. Επομένως θα πρέπει να μας τα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή τι θα γίνει με αυτό το μοναδικό μέσο. Πώς θα μπορέσουμε να δούμε το πώς αντί για ευελιξία να αποφύγουμε δηλαδή, τον έχουμε κάποιο είδους ε, εναλλακτική χρήση ε, της χρηματοδότησης για κάποια θέματα προτεραιότητας όπως η μετανάστευση. Τώρα από την ΤΕΦΚΟ ο κύριος ε, Γκριμών που έχει εμπλακεί στην σύνταξη του κειμένου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε μας δώσατε το λόγο για το σημαντικό θέμα. Είμαστε ακόμα στην αρχή της διαδρομής για το MFF. Θα είναι πολιτική η συζήτηση, αλλά επί τη βάση των προτασιών μας, επί τη βάση της απόφασης της Δευτέρας Μαΐου μπορούμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα και να καταλάβουμε ερωτήσεις, προβληματισμό. Θα συνεχιστεί η συζήτηση και τον ε, Ιούνιο και έχουμε διάφορα στοιχεία σημαντικά τα οποία έχει προτείνει η Επιτροπή. που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικά για την συνεργασία. Έχουμε 26% ονομαστική αύξηση για τη χρηματοδότηση. Και έχει δίκιο ο συνάδελφος από το Κονκόρτ όσον αφορά αυτήν την αύξηση που είναι σημαντική. Τώρα, έχουμε αυτό το καινούργιο MFF των 27 και τώρα έχουμε το κεφαλαίο 4 και το Ταμείο Ανάπτυξης. Οπότε εδώ έχουμε την σημαντική αύξηση βλέπετε πώς έχουμε κορυφαία προτεραιότητα της δαπάνης για την ανάπτυξη. Εξωστρεφής είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως βλέπουμε τα πράγματα. Βεβαίως και ε, η τελική απόφαση θα ληφθεί από εσά και το Συμβούλιο αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο το ότι είναι εξωστρεφής η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτές μας τις προτάσεις όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία. Άρα θα πετύχουμε τους ποιοτικού μας στόχους. Θα πετύχουμε το 0,7% όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. είναι και θα παραμείνουν οι πόροι που προβλέπονται για την επιστημική βοήθεια και άρα θα τηρήσουμε τη δέσμευσή μας για αυτόν τον συλλογικό στόχο και τα κρατημέρια θα επίσης θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την ε, ε, ε ανάπτυξη της γειτονιάς σας περιοχής θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται και στην παγκόσμια σκηνή και θα πρέπει το θεματολόγιο του 2030 να βοηθηθεί. Πολύ θετικά τα όσα ακούσαν πλευράς Concord. Αλλά υπάρχει πρόβλημα εσωτερική συνέπεια, γιατί λέει ότι αυτό είναι ένα σημαντικό μέσο και μετά λέει ότι είναι χωριστό. Δηλαδή λέει ότι είναι μοναδικό αλλά μετά λέω ότι είναι χωριστό για την πολιτική γειτονία σα. δημοκρατία είναι στην καρδιά της πολιτικής μας. Γιατί να έχουμε χωριστό μέσο. Έτσι ε, διασπάται ο ενιός χαρακτήρας των στόχων της ε, ανάπτυξης. Έτσι η ανάπτυξη χάνει τον κεντρικό της ρόλο. να σταματήσει επομένω να υπάρχει κατάτμιση πολυφωνία στα μέσα χρηματοδότησης θα πρέπει να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία όσον αφορά την υποπτία και τη διαχείριση υπάρχει πολυνομία είναι περίπλοκο το καθεστώς και έτσι οι δικαιούχες χώρες να ωφεληθούν να γιατί αυτό το ευρύ μέσον θα ωφελείς και θα έχει θετικέ επιπτώσεις και για τις χώρες που τα χρειάζονται και για τον κόσμο που το χρειάζεται. Οπότε θα πρέπει να ε, ε, συνεχίσουμε τις πολιτικές μας και έτσι να έχουμε αυτό το ευρύ μέσον το οποίο δεν σημαίνει μία μοναδική πολιτική. Χρειάζεται συνεργασία και ο μπούσουλας είναι η Ευρωπαϊκή Συνένεση, όπως διαμορφώθηκε εδώ. Προβλεψιμότητα, διαφάνεια, ιδιοποίηση από πλευράς των κρατών μελών, όλα αυτά να είναι τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας μας. Άλλο σημαντικό είναι ότι η πρόταση της Επιτροπής σημαίνει ότι θα υπάρχει αυξημένη εποπτεία και αυξημένες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό. Και εμείς προτείνουμε όλα αυτά να ενταχθούν στον προϋπολογισμό. Και έτσι η ευελιξία αυτών των μέσων να πάνε και στον προϋπολογισμό και έτσι να αντιμετωπίσουμε τις νέες προτεραιότητες για το μέλλον. Για αυτό το ταμείο. Έτσι θα προενεργήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε σε μια πενταετία πώς θα έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Το Ταμείο Ανάπτυξης θα πρέπει να καλύψει ό,τι προτεραιότητες χρειαστεί να θέσουμε για την μέλουσα περίοδο. Όσο αφορά την διακυβέρνηση και αυτά τα μέσα ε, πολιτικής και χρηματοδότησης θα πρέπει να συνοηθούμε να έχουμε αυτόν τον δομημένο διάλογο, αυτή την ανταλλαγή επιστολών, να αντιλήσουμε συμπεράσματα του έχει γίνει για το μέλλον και να δούμε πώς θα οργανώσουμε και για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο την κατάσταση οπότε θα πρέπει να έχουμε εις βάθος ανάλυση για ανταλλαγή απόψεων τον Ιούνιο. Ο Επίτροπος Μίμητσα θα έρθει και θα σας εξηγήσει καλύτερα από μένα. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά προσπάθησα να σας εξηγήσω το πνεύμα των προτάσεών μας η Πρόεδρος. Ευχαριστώ, αλλά δεν σαν έχω κι εγώ προς εσένα κάποιες ερωτήσεις. Να δούμε τα αριθμητικά στοιχεία. Και είχαμε αυτό το σημείο με τα ποσά που έφτιαξε η Επιτροπή και διανεμήθηκε Τελικά το κριτήριο της κατανομής είναι γεωγραφικό. Ας πούμε θα υπάρχει ε, ένα ποσό, ένα κουμπαράς για την Αφρική και όχι για όλη την ανάπτυξη. Ισχύει αυτό ή πάμε πάλι στην ε, κατανομή στο κριτήριο της ε, γειτονιάς περιοχής. Αφρική, υποσαχάρη Αφρική δηλαδή. Είναι γεωγραφικό το κριτήριο και βάζουμε μέσα όλη την Αφρική. Είναι διαφορετικό αυτό. Επίσης τα έχουμε ξανασυζητήσει με συναδέλφους από την ΔΕΦΚΟ για το πώς θα πάμε για το Άντις. Για το πώς θα κάνουμε αυτά που σχεδιάζουμε προ τι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε και τι υπάρχει στο πολιτέ πλαίσιο, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε του πόρου για εκείνε τι χώρε. Προβλέπετε τίποτα στο MFF. Είπατε πάρα πολλοί από αυτούς τους πόρους είναι ε, αναπτυξιακή βοήθεια σύμφωνα με τον ΤΑΚ Δεν θέλω να στριμώξουμε κανέναν, αλλά δεν έχω καταλάβει. Τι λέει η ΕΚΟ. Καλά να μας τα πει ο Επίτροπος το απόγευμα. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα της ΔΕΒΚΟ, αλλά είναι και της ΕΚΟ. και θα σας ξαναδώσουμε το λόγο, αλλά να απαντήσει πρώτα ο Βένσα που είναι ο άμεσα αρμόδιος. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, όχι. Πες μας τα εσύ πρώτα Βενσα και μετά τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Πολύ σημαντικές, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω συγκεκριμένα σήμερα. Να, περιμένουμε. Και όπως είπαμε σαν ανακοίνωση του Μάια, να έχουμε κουμπαράδες ούτως επίν με γεωγραφικά κριτήρια και αυτή είναι η αρχιτεκτονική του χρηματοδοτικού μέσου. Είπαμε είναι ευρέως χαρακτήρος αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Ε, οπότε το θέμα αυτών των ευάλωτων χωρών και των λιγότερων επιμένων χωρών, αυτό είναι πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσουμε. Και βέβαια για το ότι θα ισχύσει το ΝΤΑΚ Α, ακόμα επομένως δεν ξέρετε, να περιμένουμε. Ε, δεν μπορεί, αφού δημοσιοποίησε την πρότασή της, θα ξέρει η Κομισιόν. Και τι γίνεται με το μέσο ευελιξία. Έμεινε 20%, πολλά λεφτά δηλαδή. Και θα γίνει έλεγχος από κοινοβούλιο, συμβούλιο. Ναι, η ευελιξία έχει πολλές πτυχές. Και από το EDF είπαμε ότι υπάρχουν κάποια κονδύλια όταν δεν έχουν απορροφηθεί πάνε σε νέες προτεραιότητες, σε νέες συνθήκες. Και ο, είπαμε ότι το Ταμείο θα πάει στον προπολισμό, αυτό είναι ε, καλά μαντάτα από πλευράς της διαφάνειας. Οπότε, έχουμε τις προτάσεις μας για τα ποσά και θα ισχύσει ως διαδικασία, ως τρόπος λειτουργίας ό,τι ισχύει ήδη για το EDF. Η σημερινή πρακτική είναι να ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες για αυτά τα κονδύλια. Γιατί να υπάρχει άλλου είδους διαδικασία λήψης αποφάσεων να δούμε ποια θα είναι η νομοθετική πρόταση. Ωραία, δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις από συναδέλφους, αλλά τον Ιούνιο όταν θα δούμε τα μέσα, νομίζω πως θα υπάρχουν και περισσότερες ερωτήσεις. Θα δώσω τώρα το λόγο στους προσκεκλημένους, πρώτα στον Ραφάηλ και μετά στην Κατραζινά. Ευχαριστώ. Εντάξει, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για την εξωτερική διάσταση. Θα ήθελα όμως να αντιδράσω σε αυτά που είπε ο κύριος Γκέρεντς. Αν σας κατάλαβα καλά, εκφράσατε κάποιες αμφιβολίες για την ε, πρόθεση να δοθεί προτεραιότητα στο περιβάλλον, στο κλίμα. Να επαναλάβω μόνο τα λόγια του Προέδρου Μακρόν όταν ε, ήταν στις Ηνωμένε Πολιτείες, πως δεν υπάρχει ε, εφεδρικό σχέδιο. Η καλύτερη πολιτική είναι να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, έτσι ώστε να μην ε, χρειάζεται ακόμα περισσότεροι άνθρωποι να μεταναστέψουν. Και χρειάζεται επίσης οι πολιτικές μας ε, να είναι ε, όλες συνδεδεμένες και να έχουν εξωτερική διάσταση. Τώρα, σίγουρα αυτή είναι μόνο η αρχή της συζήτησης, ε, όμως νομίζω πως ε, τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θα πρέπει να δείξουν περισσότερη φιλοδοξία. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο για την αύξηση αυτής της ε, φιλοδοξίας του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης, δεδομένου μάλιστα ότι προτού η Επιτροπή δημοσιεύσει στις 2 Μαΐου την έκθεση, ήδη υπήρχαν κάποια προσχέδια τα οποία ήταν περισσότερο φιλόδοξα από αυτό που είδαμε. Με συγκεκριμένα κονδύλια για συγκεκριμένους στόχους. Γι' αυτό λοιπόν θα δούμε ε, τι θα κάνει η πρόταση αυτή. Ελπίζω να βοηθήσει να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ας μην ξεχνάμε όχι μόνο όμως τους ε, πρόσφυγες αλλά και τις ε, συγκρούσεις. Αν δείτε ε, τις ε, μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές θα παρατηρήσετε ότι είναι άμεσα συνδεδεμένες με ε, τις περιοχές που παρατηρούνται ενόπλες συγκρούσεις. κυρία Λασάνισκα, έχει το λόγο. Σε ό,τι αφορά το κλίμα, ίσως κάποιοι παρόντες ξέρουν καλύτερα από μένα. Σκοπός είναι δεν είναι ε, να ε, υπάρξουν ε, περισσότερη χρηματοδότηση εκ των υστέρων, αλλά και η πρόληψη είναι πολύ σημαντική, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αιτίες των αδυναμιών, των εκτοπισμών, των πληθυσμών και όπως, και όπως είπε η κυρία Μακέβαν, των επιπτώσεων των συγκρούσεων και επίσης πρέπει να υπάρξει περαιτέρω ιεράρχηση, περισσότερες φιλοδοξίες. Αυτό τι σημαίνει, ότι χρειαζόμαστε περισσότερες δράσεις σχετικές με το κλίμα και την βιοπικιλότητα. Και ξέρω ότι κάποιοι ενδιαφέρονται για την υγεία. Σε αυτό το τομέα υπάρχουν ε, πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες, για παράδειγμα στο Lancet αν δεν αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, αν δεν παρέμβουμε για να ε, ε, αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, όσα έχουμε κερδίσει τα τελευταία 20 χρόνια στο, τελευταία, τομέα της υγείας θα ε, χαθούν. Ε, για να ενισχύσουμε λοιπόν το σύστημα υγείας πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε την απαραίτητη πρόοδο στο μέτωπο του κλίματος και σε ό,τι αφορά τον, ε, την επισητιστική ασφάλεια. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε διάφορα περιβαλλοντικά ε, προβλήματα, την όξυνση των υδάτων, των ωκεανών. Και όπως είπατε προηγουμένως πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ε, οι δράσεις που εντάσσονται στην ε, αναπτυξιακή πολιτική δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις ε, για το κλίμα ή στο τομέα της γεωργίας. Επίσης, θα συνεχίσω στα αγγλικά για να απαντήσω στην Κομισιόν. Όπως είπαμε, συνειδητοποιούμε απόλυτα ότι ο προπολογισμό αυτός είναι πολύ φιλόδοξος. Εμείς όμως αυτό που θα θέλαμε είναι να υπάρξει διασφάλιση ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα ε, προσανατολιστεί, θα λειτουργήσει, θα δομηθεί με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη. Και με βάση την πρόταση που δημοσιεύθηκε στις 2 Μαΐου, δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Η έκθεση ε, εστιάζει στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιμετώπιση της φτώχειας σε τρίτες χώρες μπορεί να αποτελέσει προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς όμως το ενιαίο χρηματοδοτικό εργαλείο που προτείνεται είναι πολύ ευρύτερο από την ε, καθ' αυτή αναπτυξιακή πολιτική. Υπάρχουν εντάσεις που δεν αντιμετωπίζονται. Ε, αυτά μας απασχολούν και επίσης. Ε, φοβόμαστε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια θα υπονομευτεί αν ενταχθεί σε άλλους στόχους και η μετανάστευση είναι ε, παράδειγμα. Το είδαμε η μετανάστευση έχει ε, λάβει ε, προτερότητα απέναντι στην ανάπτυξη. Όταν κοιτάμε λοιπόν το νέο καταπιστευματικό ταμείο, ε, εντάξει, έχουν, έχουμε πολλά τέτοια ταμεία. Στόχος είναι να ενισχυθεί η ευελιξία, όμως ε, δεν είναι ε, η καλύτερη προσέγγιση να εστιάσουμε αποκλειστικά στην μετανάστευση. Αυτό πιστεύουν και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μία όθηση στην αποτελεσματικότητα των, ε, της ε, αναπτυξιακής βοήθειας. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση ναι να έχει ε, στο νου της τα δικά της συμφέροντα αλλά και τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής. Και δεν νομίζω παρόλα αυτά ότι είναι αντιφατικές οι θέσεις μας συνεχίσουμε τις συζητήσεις βέβαια και σε ό,τι αφορά την, ε, το εργαλείο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το εργαλείο για την ε, σταθερότητα και την ειρήνη. Συμφωνούμε με τις απόψεις ε, που έχουν εκφραστεί από τα δύο μεγαλύτερα δίκτυα σε αυτούς τους τομείς. Και αυτά τα δύο δίκτυα ζητούν διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία που να ε, διασφαλίζουν τις διακρίσεις. Με τα νέα, το νέο εργαλείο που προτείνεται πρέπει να ε, δούμε αν θα διασφαλιστεί η απαραίτητη διάκριση. Η συζήτηση είναι ανοιχτή. Όπως και να αν υπάρχει ένα εργαλείο για την εξωτερική πολιτική και ένα εργαλείο με πολλαπλούς στόχους που εντάσσεται στη διμερή συνεργασία, το πιθανό είναι στο μέλλον κάποιοι στόχοι αναψιακής πολιτικής να μην ληφθούν επαρκώς υπόψη. Αν υπάρχουν ταυτόχρονες διαπραγματεύσεις για διάφορους ε, στόχους και προτεραιότητες, θα δοθεί η απαραίτητη σημασία στους ε, ε, στόχους που αποτελούν προτεραιότητα. Γι' αυτό δεν είμαστε εντελώς πεπισμένοι ότι υπάρχουν οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ήθελα να ε, ε, υπάρξει λάθος κατανόηση σε ό,τι αφορά την σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Τα κράτη-μέλη ε, δεσμεύονται ε, στον τομέα της χρηματοδότησης και μετά δεν ε, τις τηρούν. Δεσμεύσεις στα πλαίσια της COP21 και μετά δεν τις τηρούν. Ε, υπόσχονται τεράστια ποσά στις αναπτυσσόμενες χώρες για να διορθωθούν τα λάθη του παρελθόντων και δεν τις τηρούν. Δεν τηρούν τις δεσμεύσεις που ε, ανακοινώνουν στις μεγάλες ε, διεθνείς ε, διασκέψεις και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Συμφωνούν με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, δεν καθορίζουν όμως τη μέθοδο επίλυσης των προβλημάτων. Δεν υπάρχει μέθοδος, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το τι θα κάνουν μέχρι το 2030 η έκθεση στέλνει σαν να μην υπήρξε ε, ποτέ, παρόλο που καλεί όλους να αναλάβουν τις ε, ευθύνες τους. Εγώ αυτό που διαπιστώνω είναι το εξής. Όλοι εστιάζουν στην ε, Κομισιόν που έχει υπό τον έλεγχο της, τα ποσά, τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου ε, ανάπτυξης. Αλλά τα κράτη-μέλη τι κάνουν. Τα κράτη-μέλη που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους ουσιαστικά ε, συμφωνούν παράλληλα ταυτόχρονα με την Κομισιόν τι ποσά θα διατεθούν σε τι ε, δράσεις. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Και φοβάμαι ότι το ποσό που έχει στη διάθεσή της ε, η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση ε, κινδυνεύει να διατεθεί για τη διόρθωση λαθών του παρελθόντος χωρίς να είμαστε επαρκώς στρεμμένοι προς το μέλλον. Γι' αυτό δεν είμαι υπέρ της χρηματοδότησης των δράσεων για την κλιματική αλλαγή. Άλλοι τομείς χρειάζονται ενίσχυση των πόρων. Δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο ένα πολύ μικρό ε, κομμάτι όλων των πολιτικών που καλείται να υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό και είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί ε, των ε, δράσεων και στον τομέα ε, του περιβάλλοντος και στο τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση έχω ακόμα, Φανσά. Προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, πήγαμε στην ουγγάντα την περασμένη εβδομάδα και είδαμε ότι ένα από τα προβλήματα είναι η χρηματοδότηση αυτού του συνδέσμου. Προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε τα καταπιστεύματα για την χρηματοδότηση, μακροπρόθεσμα. Ε, προτίθεστε λοιπόν να χρηματοδοτήσετε μακροπρόθεσμα έργα ε, σχετικά με το προσφυγικό. Δεν ξέρω πώς φαντάζεστε ότι θα διαχειριστείτε στην πράξη τα προγράμματα αυτά. Έχουν ήδη διαπιστωθεί προβλήματα στο πρόγραμμα που τρέχει για αυτήν την επταετή περίοδο. Τα καταπιστεύματα που έχουμε δημιουργήσει, το τα δημιουργήσαμε επειδή ακριβώς μας έλειπε η ευελιξία. Γι' αυτό λοιπόν θα χρηματοδοτηθεί αυτός ο ε, σύνδεσμος ε, για μακροπρόθεσμα προγράμματα που θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση ε, εκτεταμένων κρίσεων. Γιατί στην Ουγκάντα το είδαμε ότι τα κονδύλια κατανέμονται ετησίως σε συγκεκριμένα έργα. Και σίγουρα κάποιες κυβερνήσεις είναι περισσότερο πρόθυμες από άλλες για να αναλάβουν δράσεις. Όταν λαμβάνουν κονδύλια, τότε ορισμένε κυβερνήσει εστιάζουν ε, στι δικέ του προβληματικέ περιοχέ και δεν βλέπουν το γενικότερο πλαίσιο. Έχετε λοιπόν σκεφτεί τι ε, λεπτομέρειε στην πράξη, τα προβλήματα. Θα υπάρχει ουσιαστική ε, εταιρική σχέση με τις χώρες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το σκεπτικό πίσω από την πρόταση είναι να προσπαθήσουμε να ε, έχουμε μία από τις ε, καλύτερες ε, δυνατές πρακτικές και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αυτού. Τώρα σε ό,τι αφορά του, τις διάφορες συνδέσεις υπάρχει ένα ευρύτερο μέσο γενικότερο θα είναι χαρακτηρισμό καινοτομία, θα διαθέτει δικό του κονδύλι προϋπολογισμού για την ανάπτυξη. Θα υπάρχει αυτό που λέμε δημιουργία ανθεκτικότητας και θα φροντίσουμε να καλύψουμε τα κενά. Διότι αυτά είναι θέματα που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει έρθει όμως η ώρα να τα υλοποιήσουμε. Η καινοτομία λοιπόν είναι κέρια σημασίας για να στηρίξουμε αυτόν τον σύνδεσμο. Και σίγουρα η συζήτηση θα πρέπει να συνεχιστεί στο πλαίσιο του σχεδίου κανονισμού, διότι πρόκειται για νομικό ακριβώς κείμενο, το οποίο δεν έχει όμως ακόμα εγκριθεί. Να τονίσω όμως δύο πράγματα. Πρόθεσή μας είναι το μέσο αυτό να καλύπτει και την ε, πολιτική γειτονίας και σήμερα τα ενωσιακά προγράμματα είναι ως επιτοπλίστων ε, για επίσημα αναπτυξιακή βοήθεια. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε τις ε, λεπτομέρειες. Σίγουρα υπάρχουν έτσι, διαφορές στα επιμέρους όμως όλα υπάγονται στην επίσημα αναπτυξιακή βοήθεια. <coughs> Υπάρχει λοιπόν δυναμικό για τη δημιουργία ενός μέσου που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Ε, διότι αν συνεχίσει η κατάσταση έτσι όπως είναι, πολύ φοβάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορεί να τηρήσει τις υποσχέσεις της. Πράγματι, γιατί ακούσαμε και από άτομα που είναι εκεί επιτόπου πως έχουν τα ίδια προβλήματα με τις ε, περασμένες χρονιές, ότι τους έχουν στερέψει τα κονδύλια δεν μπορούν να προγραμματίσουν τους επόμενους ε, μήνες, γιατί ακριβώς τα κονδύλια έρχονται με δόσεις. Χρειάζεται πολυετής προγραμματισμός και όπως ε, ακούμε πολλές φορές καλά τα λόγια, αλλά ας περάσουμε στις πράξεις. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα κάθε χρονιά και να ε, ψάχνουμε να βρούμε τα επόμενα κονδύλια για το μέλλον. Τώρα πρέπει να γίνουν αυτά. Όπως είπατε όμως και εσείς υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία προς το παρόν παραμένουν αναπάντητα. Τι σημαίνει γειτονία, τι σημαίνει Αφρική, τι σημαίνει αναπτυξιακή βοήθεια. Νομίζω πως ε, μέχρι τον Ιούνιο όμως ε, θα πρέπει να μας ε, δώσετε κάποιες απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Θα συνεχίσουμε την συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Okay, colleagues. Συνάδελφοι, σε δύο λεπτά θα έρθουν και οι προσκεκλημένοι για το θέμα για το Σουδάν, οπότε διακόπτουμε μέχρι τις 12 παρατέταρτο. Και μην ξεχνάτε 12 και 4 ψηφίζουμε.

Okay, colleagues, our guest speakers have arrived here. Ήρθαν εδώ οι προσκεκλημένοι μας ομιλητές. Ε, και στην γαλαρία, παρακαλώ, αν θέλετε να τα πείτε, περάστε έξω. Και προχωρούμε τώρα στο θέμα υπαριθμών εννέα. Και έχουμε εδώ τους καλεσμένους μας που θα μας μιλήσουν, που καθυστέρησαν στο Συμβούλιο. Δυσκολεύτηκαν, πέρασε ώρα για να τους αφήσουν να μπουν και καθυστέρησαν στο Συμβούλιο αλλά ήρθαν και θα συζητήσουμε ε, για το Σούδαν το ανθρωπιστικό σε σχέση με την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους πιο βασικούς ε, δωρητές για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη χώρα. Και ξέρετε μόλις ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για το πολιτές δημιουργικό πλαίσιο, τα είπαμε και στο γραφείο μου για την μακρόπνη βοήθεια, την ανθρωπιστική βοήθεια και για αυτή την πολιετή χρηματοδότηση πήγαμε στην Ουγκάντα και εκεί οι συνάδελφοι μου είπαν ότι όλη τους την ζωή αντί να δουλεύουν επί τόπου ασχολούνται με τις συμβάσεις η μία ακολουθεί την άλλη Τα απόγευμα πάντως θα μιλήσουμε με τους ε, επιτρόπους με την Επιτροπή γενικότερα οπότε θέλουμε να μας τα πείτε όλα Πώς θα οργανωθεί το νέο πρόγραμμα. Έχει προτεραιότητα η χώρα σας, πήγαμε και στην, ε, στην Ουγκάντα. Ξέρουμε ότι τα προβλήματα στη μία χώρα συνδέονται με την άλλη. Πολύ σημαντικό να υπάρχει ασφάλεια στο Σουδάν. έχουμε τον κύριο Χόλιγουρθ, έχουμε την κυρία Μακουάνα ε, από το Γραφείο Συντονισμού και θα τους δώσουμε τον λόγο. Ο πρώτος κύριος είναι από το Παγκόσμιο Πιστητικό Πρόγραμμα. 12 και 4 θα πρέπει να ψηφίσουμε οπότε έχετε ένα πεντάλεπτο ο καθένας Χόλιγκουρτ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους βουλευτές μας καλέσατε σήμερα για να συζητήσουμε για κάποια πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα το Σουδάν όπως γνωρίζετε ε, εδώ και 15 χρόνια και παραπάνω υπάρχει πρόβλημα στη χώρα, υπάρχει εμφύλιος ε, πόλεμος, ο ένας Σουδανός πόλεμα τον άλλο. Και το 2011 αποσχίστηκε τον με της χώρας και από τότε έχουμε αργή αλλά σταθερή επιδείνωση της ε, οικονομίας. Οπότε τώρα έχουμε δύο χώρες δέχθηκε το Σουδάν, το χρέος του Νότιου Σουδάν και τα τελευταία πενταετία η επιδείνωση επιταχύνθηκε και αρχάς του 18 λόγω του ότι υπήρχε έλλειψη αποθεματικού σκληρών νομισμάτων δεν μπορούσε η χώρα να πληρώσει τις εισαγωγές δεν μπορούσε να συνεχίσουν τις ε, ενισχύσεις προς ε, βασικά εμπορεύματα για τρόφιμα, για καύσιμα και είδαμε ότι διπλασιάστηκε η τιμή του ψωμιού και τέτραπλασιάστηκε η τιμή του σόργου ε, και άλλων ε, προϊόντων. Το ίδιο και όσον αφορά τα διελιστήρια καυσίμων και όταν δεν υπάρχουν ε, καύσιμα δεν μπορούν να κινηθούν τα φορτηγά, δεν μπορούν να μεταφερθούν τα εμπορεύματα και το φαγητό γύρω γύρω στη χώρα. Έχουμε τώρα 55% πληθωρισμό με ανωδικές τάσεις και παραδοσιακά εμείς σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους εκτοπισμένους από τον εμφύλιο πόλεμο, να υποστηρίξουμε τους πρόσφυγες από τον Νότιο Σουδάν, 1,2 εκατομμύρια είναι αυτοί και 800.000 είναι από τον εμφύλιο στο Νότιο Σουδάν, οπότε όλοι αυτοί που παρασυγά τους βοηθούμε ε, κατά 98-99% δεν μπορούν να βρουν τα προς το ζήν κάθε μέρα τα τρόφιμα που χρειάζονται για να μην μιλήσουμε για παιδεία και ε, ιατρικές ε, φροντίδες. Δυστυχώς τώρα πάρα πολλοί από αυτούς που είχαν εκτοπιστεί αρχές δεκαετίας του 2000 τώρα επιστρέφουν αλλά και αυτοί είναι πολύ ευάλωτοι και αυτοί θέλουν πιστιστική βοήθεια και άλλα είδη βοήθειας οπότε για πρώτη φορά βλέπουμε σε πάρα πολλά μέρη κάποιοι που δεν έχουν φυγεί από τον εμφύλιο αυτοί ενώ έχουν δουλειά, ενώ έχουν ένα χωράφι δεν μπορούν να καλύψουν τις ε, ανάγκες τους λόγω της κρίσης που σοβεί στη χώρα. Είπαμε αύξηση των τιμών και ανεπάρκεια προσφοράς. Οπότε ακόμα και αν κάποιο βρει τα λεφτά δεν μπορεί να βρει τα προϊόντα, τα απαραίτητα. Οπότε όλα είναι και πιο δύσκολη κατάσταση στη χώρα προβληματιζόμαστε βαθύτατα. Έχει επτά γειτονιάρουσες χώρες το Σουδάν και όλες αυτές οι χώρες ε, χαρακτηρίζονται ευάλωτες. 42 εκατομμύρια είναι ο πληθυσμός της χώρας και 230 εκατομμύρια ο πληθυσμός ε, ο ευάλωτος πληθυσμός αυτών των 7 γειτόνων. Η χώρα από κάπως σταθεροποιούσε, τώρα και αυτή όλο ένα γίνεται πιο ασταθής και όλο ένα και περισσότεροι εκτοπίζονται. Όλο ένα και περισσότεροι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν λόγω αυτής της κατάστασης. Επίσης, η αποστολή μας στο Νταρφούρ, στο Ιουνμίτ τώρα αποσύρεται βαθμία σε δύο χρόνια. Θα φύγουν από τον Νταρφούρ και αυτό και για θετικούς λόγους γιατί ισχύει η κατάβαση πυρός, υπάρχει η ειρήνη ε, τώρα με τα 15 χρόνια και γι' αυτό αποφασίστηκε η σχετική ταχεία α, ε, αναχώρηση της UNMID. Πάντως ε, το πρόβλημα είναι ότι με το που θα φύγει η δύναμη θα πρέπει να συνοδευτεί από το να ειρηνεύσει περισσότερο το δυτικό τμήμα της χώρας. Περίπλοκη, δύσκολη χώρα. Συνεχίζει να περτοδούμε τον Μπασίρ, τον πρόεδρο Μπασίρ. Το Σουδάν συνεχίζει να θεωρείται ότι βοηθά την τρομοκρατία από τη ΣΥΠΑ δισεκατομμύρια ε, δολαρίων χρέος, προσφεύγουν στο Λέσχο των Παρισίων, στην Κοτονού. Όλα αυτά σημαίνουν ότι δάνεια και αναπτυξιακή βοήθεια δεν έρχεται και δεν μπορεί να έρθει. Δεν μπορεί το σύστημα να λειτουργήσει. Η ανθρωπιστική βοήθεια από Αμερική, Αγγλία και Ευρώ βοηθά, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα δολάρια που θα έπρεπε να έρχονται για ειρήνευση και ανάπτυξη. Άρα το πρόβλημα επιδεινώνεται. Επιτεύχθη πρόοδος όταν το Σουτάν θεωρήθηκε πιλωτική χώρα για αυτή τη σύνδεση ανθρωπιστικής βοήθειας με την ανάπτυξη βοήθεια, ανάπτυξη και ειρήνευση ήταν οι τρεις πυλώνες αυτού του προγράμματος. Οπότε μέσω των απόψεων των χωρών μελών προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον προγραμματισμό μας και κάτι που το οποίο θα ωφελήσει τη χώρα. Βελτίωση όσον αφορά την εμπλοκή της κυβέρνησης για να μπορέσουν να είναι υπόλογοι σε σχέση με το τι έχουν υποσχεθεί ως κυβέρνηση για τον λαό τους να συντονιστούν μαζί μας οπότε έχουμε κάποια βήματα πρόοδου σε αυτό το μέτωπο όμως αυτό το οποίο δεν γίνεται είναι αυτό που είπε η πρόεδρος δεν βλέπουμε την πολυετή χρηματοδότηση που χρειαζόμαστε την ευέλικτη χρηματοδότηση που χρειάζεται για όλα αυτά τα οποία είπαμε τις, αυτές τις συνδεδεμένες ε, ανάγκες ανθρωπιστικό, ανάπτυξη κλπ. Έχουμε 7,1 εκατομμύριο πρόσωπα τώρα που χρειάζονται βοήθεια και, και άλλα 42 που έχει η χώρα. Όλοι αυτοί θα ωφελούνται αν υπήρχε η αρρωγή. Έχουμε ακόμα 4 εκατομμύρια δολάρια που χρειάζονται και δεν τα έχουμε όλα. Μόνο ένα κλάσμα αυτό που χρειάζεται για την ανθρωπιστική βοήθεια. Οπότε η ανάγκη φέρνει αστάθεια, πολιτικά προβλήματα, προβλήματα στην καθημερινή ζωή. Δεν μπορεί ο κόσμος να βγάλει το ψωμί του, να σταροποιήσει τη ζωή του. Επομένως είναι ευάλωτη η όλη περιοχή και αν ε, εκραγεί το Σουδάν όλοι θα θυγούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρωτού δώσω το λόγο στα μέλη, αναφερθήκατε σε υπουργούς, πήγατε δηλαδή στο Συμβούλιο. Ε, τι ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, Ας συζητήσουμε το θέμα της ε, προσέγγισης της ανθρωπιστικής βοήθειας στην ενευτική διαδικασία. Ας ε, δούμε πώς ε, μπορούμε να παρέχουμε πολυετή ευέλικτη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ας δούμε πώς μπορούμε να σκεφτούμε εκτός πλαισίου έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι το Σουδάν δεν θα αποστεθεροποιηθεί σε σημείο που θα έχουμε όλο τον πληθυσμό του να ψάχνει ασφάλεια και ε, εκτός της χώρας. Ναι, πριν αναφερθήκαμε σύντομα στο Κονγκό και τον ε, κίνδυνο κατάρρευσης της χώρας και πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά για πλήθη προσφύγων από την ε, χώρα αυτή. Αλλά υπάρχουν ε, εκατομμύρια εκτοπισμένοι και στο Σουδάν, ε, προς τον Νότιο Σουδάν, προς την Ουγγάντα. Αυτό είναι δοκιμασία για τον μηχανισμό πρόληψης ανθρωπιστικών καταστροφών. Όμως όπως ε, συνήθως βλέπουμε ελάχιστα κονδύλια. Να ε, σας ε, ρωτήσω πώς ακριβώς είναι τα χρήματα. 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι λιγότερο από το 1 τέταρτο του, των χρημάτων που χρειάζονται. Η Σεσίλ Κιέγγι έχει να σας κάνει μια ερώτηση. Συμπάθετε με γιατί είχα κάποια υποχρέωση και άργησα να έρθω, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό το πόσο επήγει η κατάσταση στην, στον στον και τι γίνεται στο Σουδάν. Ε, πολλές φορές να φύγουν και να, να, να περάσουν μέσω Νίγηρα, να πάνε στην ε, Λιβύη ε, και ο Νίκηρας τώρα όμως ε, έχει πρόβλημα όσον αφορά τους Σουδανούς που καταφεύγουν εκεί. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ωραία, ας απαντηθεί αυτή πρώτα. Λοιπόν, σίγουρα όλη η περιοχή του Σαχέλ έχει προβλήματα. Και υπάρχουν μετακινήσεις πληθυσμών στην υποσαχάρια Αφρική, οι οποίοι ψάχνουν τρόπο να πάνε πιο βόρεια. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το Σουδάν είναι πύλη προς τη Λιβύη και μέσω αυτής πύλη προς την Ευρώπη. Και ακριβώς όπως έχουν ε, μετακινηθεί εκτός Σουδάν οι Σουδανέζοι για να βρουν ασφαλέστερες συνθήκες, όπως σας είπα υπάρχουν 2,8 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Αιθιοπία, την Ερυθρέα, το Τσάντ, κυρίως από τον Νότιο Σουδάν αλλά υπάρχει και αυξανόμενος αριθμός ε, σύρων. Το Σουδάν ανοίγει τις πόρτες του στους πρόσφυγες και τους επιτρέπει να ταξιδέψουν και να εργαστούν στη χώρα ελεύθερα. Όμως ε, δεν μπορούν να δουλέψουν διότι η οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα και η κατάσταση επιδεινώνεται συνέχεια. Μειώνεται και η ανθρωπιστική βοήθεια, ακριβώς διότι μειώνονται τα κονδύλια και δεν θα μπορούν οι πρόσφυγες αυτοί να παραμείνουν εκεί για πολύ καιρό. Ε, όπως γνωρίζω, έχει πετρέλαιο το Σουδάν, στο νότιο Σουδάν αν δεν κάνω λάθο, Θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό. Δεν υπήρχαν ε, πολλές συνδέσεις με την Κίνα, αν γνωρίζω καλά. Το 2009 θυμάμαι στην ε, Κοπενχάγη το Σουδάν είχε ηγετικό ρόλο στην, ε, ανάμεσα στις χώρες της ε, Αφρικής και μάλιστα εμπόδιζε τις εξελίξεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τι γίνεται λοιπόν με το πετρέλαιο στο Σουδάν, με τα χρήματα που αποφέρει η εξόριξη πετρελαίου και τι γίνεται με την συνεργασία από την κυβέρνηση. Μας είπατε για την κυβέρνηση Μπασίρ δεν ξέρω τι γίνεται, αναφερθήκατε στο Διεθνές Δικαστήριο. Πώς μπορείς να δουλέψει, να εργαστείς σε μια χώρα όπου η κυβέρνηση αρνείται να συνεργαστεί. Διότι φαντάζομαι ότι από τη δική τους ε, πλευρά θεωρούν πως ε, η παγκόσμια κοινότητα τους ε, πολεμούσε γιατί προσπαθούσε να βοηθήσει την ανεξαρτητοποίηση του Νότιου Σουδάν. Τι θα έχετε λοιπόν να πείτε γι' αυτό. Πολλές και καλές ερωτήσεις σας. Πρώτον, η συντριπτική πλειοψηφία των κοιτασμάτων πετρελαίου βρίσκεται στο νότιο Σουδάν. Και όταν είχε παρατηρηθεί άνθηση της οικονομίας μέχρι τη διάσπαση της χώρας, τότε το νότιο Σουδάν εξόρισε πετρέλαιο, γινόταν η δίληση στο Σουδάν και μετά ε, εξαγόταν αυτό στις υπόλοιπες χώρες. Αυτό όμως σταμάτησε και αυτό σημαίνει πως ε, σταμάτησαν και τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου. Οι κινέζικες επενδύσεις στο Σουδάν αφορούν κυρίως εξορυκτικές δραστηριότητες, όχι μόνο πετρελαίου αλλά και χρυσού, γιατί υπάρχουν κοιτάσματα χρυσού στη χώρα. Αυτές οι επενδύσεις όμως ε, μειώνονται ακριβώς διότι η χώρα έχει χρεοκοπήσει και τα στοιχεία αυτά μας τα δίνουν ε, έγκυρες πηγές όπως η Παγκόσμια Τράπεζα. Δεν υπάρχουν λοιπόν λεφτά στο Σουδάν. Έπειτα, Σίγουρα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, διότι σε δύσκολους καιρούς οι κυβερνήσεις ε, παρατηρείται ότι είναι πιο δεκτικές στη συνεργασία. Για άλλους ε, ίσως λόγους, όμως η αλήθεια είναι αυτή. Προσπαθούν λοιπόν ε, να συνάψουν εταιρικέ σχέσεις με τις άλλες χώρες. Για να το κάνουν όμως αυτό πρέπει να παραδεχτούν ότι χρειάζεται να συνεργαστούν και να αποδεχτούν κάποιες από τις προϋποθέσεις που θέτουμε για τη συνεργασία αυτή. Και το γραφείο ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι διεθνεί οργανισμοί μαζί με την Ένωση προσπάθησαν να συγκεντρώσουν πόρους σε ένα ταμείο για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Με σκοπό να προσπαθήσουν να υλοποιήσουν αυτές τις πολύ δύσκολες διαρθρωτικές αλλαγές στο Σουδάν. Ε, διατίθενται 3-4 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια για αυτό το σκοπό. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν τα κονδύλια και διατεθούν, αυτό θα σημαίνει ότι τα διατεθούν υπό προϋποθέσεις και ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να σεβαστεί κάποια θεμελιώδη δικαιώματα, ελευθερίες, κράτος δικαίου και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πλαίσιο συζητήσεων, διότι ακριβώς ε, αυτό συνέβη. Η κυβέρνηση του Σουδάν έχει αναγνωρίσει πως χρειάζεται βοήθεια και έχει αναγνωρίσει πως κάπως πρέπει να ε, απελευθερώσει αυτά τα κονδύλια. Ε, κυρία Κέγκε, θα σας δώσω το λόγο μετά για να απαντήσετε, αλλά τώρα θα δώσω το λόγο στη... σε εσά. Ευχαριστώ και συμπαθέτε με γιατί δεν είχα την ακριβή απάντηση για την ερώτηση. Ίσως γιατί κάτι έλειπε από την ερώτηση. Μίλησα για το πόσο κατεπίγουσε είναι η κατάσταση όσον αφορά του Σουδανού στον Νίγηρα, εκεί όπου υπάρχει ένα πρόγραμμα που τρέχει για την ε, επανεγκατάσταση. Και ε, όμως αυτοί που καλύπτουν το πρόγραμμα δεν είναι Σουδανέζοι, είναι άλλοι λαοί. Αυτοί λοιπόν δεν είναι επιλέξιμοι και τους επαναπροωθούν στη, στις χώρες τους. Αυτοί οι άλλοι. Όμως η Σουδανία είναι πάρα πολύ και δεν κρατούνται από κανένα από τα προγράμματα που τρέχουν στον Νίγηρα. Δεν μπορώ να πω ε, συγκεκριμένα τι συμβαίνει με τους πρόσφυγες ε, από το Σουδάν στο Νίγηρα. Δεν διαχειριζόμαστε αυτό το θέμα. Μπορώ να σας πω τι συμβαίνει στην Κεντρική Αφρική, στο Τσάντ. Κάποιοι επιστρέφουν στο Σουδάν γιατί ε, η κατάσταση σε αυτές τις δύο χώρες είναι πολύ δύσκολη και αυτό οδηγεί κάποιους να επιστρέφουν ε, στο Νταρφούρ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω την κατάσταση στον Ήγυρο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, απευθύνομαι στην DG ECO είναι εδώ ο Μιχαήλ Ζούπατσικ. Θα ας ε, μιλήσετε οι ίδιοι. Εκπροσωπώ την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ ε, στο Σουδάν και στην, ε, στο Νότιο Σουδάν. Θα ήθελα να σας πω πρώτα απ' όλα ότι ως Γενική Διεύθυνση συμμεριζόμαστε αυτή την, την κατάσταση, τη ζωφερή κατάσταση που σας έχει περιγραφεί. Είναι πολύ αρνητικές ε, οι επιπτώσεις και τώρα έχουμε επιπλέον 1,6 εκατομμύρια άτομα που χρειάζονται ε, βοήθεια. Συνολικά 7 εκατομμύρια άνθρωποι το 2018 χρειάζονται αναπτυξιακή βοήθεια. Το επιπλέον κόστος ε, κόστος που έχει υπολογιστεί από τον ΟΗΕ είναι 500 ε, εκατομμύρια μέχρι τώρα. σε ό,τι αφορά τις διάφορες πρωτοβουλίες του ΟΗΕ ε, σχετικά με το σύνδεσμο μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης. Θα ήθελα να χαιρετήσω την ανάληψη αυτών των ε, πρωτοβουλειών και χαίρομαστε που είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στην υλοποίηση των δράσεων, των σχετικών δράσεων. Όπως γνωρίζετε ίσως ε, θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το Σουδάν είναι κέρια ε, χώρα για την ε, διαμόρφωση αυτή του συνδέσμου. Ε, έχουν υλοποιηθεί κάποιες δράσεις, κάτι που δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες που δυσχεραίνουν την υλοποίηση του συνολικού προγράμματος, δυσχερίες ως προς τη χρηματοδότηση το Σουδάν δεν έχει επικυρώσει την συμφωνία του Κοτονού σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια σε τίσια βάση ε, έχουμε, κατανέμουμε κονδύλια της τάξης του ενός δισεκατομμυρίου ε, ευρώ συμπληρώσαμε αυτή τη χρηματοδότηση με άλλα κονδύλια από, θέματα έκτακτης ανάγκης ή από το ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Είναι ε, περιορισμένοι οι πόροι, λοιπόν. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ανταποκριθούμε, αλλά οι ε, πόροι είναι περιορισμένοι. Το 2017 κινητοποίησαμε 46 ε, εκατομμύρια ευρώ για να προσφέρουμε αναπτυξιακή βοήθεια στο Σουδάν, κάτι που ήταν δυνατό χάρη στη μεταφορά κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και από την αξιοποίηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Ε, φέτος ξεκινάμε με 23 εκατομμύρια και θα δούμε αν μπορούν να αυξηθούν τα κονδύλια για να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες. Η κατάσταση φυσικά που σας έχει περιγραφεί είναι ε, πολύ ε, ευρύτερη, ε, μεγαλύτερη οι ανάγκες. Αυτά μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή η ΕΚΟ ε, φυσικά σας έχουν περιγραφεί πολύ ε, μεγαλύτερα ε, μακροοικονομικά προβλήματα. Αυτά με λίγα λόγια ήθελα να σας πω. Συζητήσαμε με τα κράτη-μέλη για συγκεκριμένα προγράμματα δράσης για την ολοποίηση του συνδέσμου. Συζητήσεις έλαβαν χώρα των... Απρίλιο και τους ερχόμενους ε, μήνες ε, ε, και από την πλευρά της ΕΚΟ και από την πλευρά της ΔΕΦΚΟ προβλέπεται υλοποίηση κάποιων δράσεων με κάποια μικρά κονδύλια που θα διατεθούν στο Σουδάν. Πολύ καλό παράδειγμα ε, τι σημαίνει στη πράξη ε, το να μην υπάρχει ένα πολιετές ε, πρόγραμμα χρηματοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και δεν μπορούν να υλοποιηθούν κατάλληλα προγράμματα. Δίνεται έκτακτη βοήθεια. Το είδαμε και στην Ουγκάντα. Εκεί χρησιμοποιήθηκαν κονδύλια από το καταπιστευματικό ταμείο για την αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων. Αυτό είναι ε, θέμα που πρέπει να κοιτάξει η DG ECO σε ό,τι αφορά το σύνδεσμο. Ε, αν θέλετε κάτι ε, τελευταίο να πείτε, τώρα είναι η στιγμή γιατί μετά έχουμε ψηφοφορία. Είχαμε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση και αν δεν ε, κινητοποιηθούμε τώρα η κρίση αυτή θα λάβει μεγαλύτερες ε, διαστάσεις. Ε, η ασάφεια που επικρατεί στο Σουδάν κινδυνεύει να οδηγήσει σε κατάρρευση και πρέπει να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση και πολύ φοβάμαι ότι εξαιτία της έλλειψης ε, κοντιλίων ε, θα ε, υπάρξει τεράστια έλλειψη τροφίμων το Σεπτέμβριο και η κρίση θα είναι πολύ χειρότερη. Και πράγματι πρέπει να εξετάσουμε ταυτόχρονα το θέμα των ανθρωπιστικών προβλημάτων και των πολιτικών λύσεων όταν μιλάμε για μια χώρα πρέπει πάντα να βγάζουμε ένα χάρτη, να βλέπουμε ποιες είναι οι γειτονικέ ε, χώρες και πού κατευθύνονται ε, οι πληθυσμοί που μεταναστεύουν προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και με ακροπρόθεσμα τα προβλήματα στο τομέα της ανάπτυξης. Θα ε, συζητήσουμε με τον Επίτροπο Σιλιανίδη σήμερα το απόγευμα. Σίγουρα θα συζητηθούν πολλά ε, θέματα σχετικά με αυτά που αναφέρατε. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, περνάμε στη ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας περάσουμε τώρα στο σημείο 10. Συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ιράκ. Είναι γνωμοδότηση για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο κύριο Βάρινεν είναι ο εισηγητής. Θα θέλατε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Λίγα λόγια μόνο να πω. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις τροπολογίες που υπέβαλαν. Δυστυχώς δεν υπήρχε περιθώριο συμβιβαστικών τροπολογιών, γι' αυτό οι ψηφοφορίες θα είναι χωριστές. Ε, κατάφερα να συμφωνήσω για τις περισσότερες τροπολογίες. Οι πιο πολλές από αυτές καλύπτονται έτσι και από το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Νομίζω πως ε, οι τροπολογίες είναι λίγο πολύ εξαιρετικές. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ωραία, ας κάνουμε μια δοκιμή να δούμε αν λειτουργούν όλα σωστά. Μπορείτε να πιέσετε οποιοδήποτε κουμπί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Μια χαρά λειτουργεί. Πολύ ωραία. Περνάμε στην τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά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 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 11 ψήφι κατά 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχέ 21 υπέρ κατά αποχέ 22 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται, 23 υπέρ κατά απόχέ απορρίπτεται, 24 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται, 25 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται, 26 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, 27 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 28. Καταπίπτει 28. 29. Υπέρ, κατά. 29. Άλλη μια φορά υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 29. Άρχεται η ψηφοφορία.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 Α, 21, με 21 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Και καμία αποχή. Με μεγάλη πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι, επιστρέφουμε στις 2 και μισή. Σας ευχαριστώ.